Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. Ας ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Avant de commencer notre séance. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν. Να απευθυνθώ στους Βέλγους φίλους μας και στα θύματα του ατυχήματο της Λουβέ που συνέβη στις 18 Φεβρουαρίου που μας πέρασε. Από πλευρά της συνελεύσεώς μου απευθύνω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του νέου που απεβίωσε και ειλικρινή υποστήριξη σε εκείνους που έζησαν το δράμα ή τραυματίστηκαν. Τα αίτια του δυστυχήματος είναι άγνωστα ακόμα έχουν λοιπόν ξεκινήσει έρευνες και όταν υπάρξουν πορίσματα που θα μας δημοσιοποιηθούν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε στην εφαρμογή του τέταρτου συνδρομικού πακέτου να λάβουμε υπόψη τα μαθήματα από το ατύχημα της Λουβέν. Η ασφάλεια σιδηροδρόμους, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Επιτροπή μας. Στο τρένο της Λουβέν επέβαιναν 80 άτομα και πληγώθηκαν κάποιοι. Τα συνδρομικά ατυχήματα έχουν σοβαρές συνέπειες. Η Ευρώπη θα συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης. Ξανά εκφράζω τη συμπάθειά μου προς το βελγικό λαό, την υποστήριξή μου προς το βελγικό λαό σχετικά με αυτή την τραγωδία. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει, Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και ξεκινάμε με την πρώτη συζήτηση, κοινή συζήτηση. Για την καταγραφή ατόμων που επιβαίνουν επιβατικών σκαφών. Έκθεση Bilbao, σύστημα επιθεώρησης για τις τεχνικές διασυνοριακές συγκοινωνίες, ε, οδικές συγκοινωνίες, ο κύριος Ρικέ και ικανό προδιαγραφές ασφαλείας για τα πλοία, τα επιβατικά της κυρίας Αγιούντο. Έχουμε πολύ φορτωμένη σε διάταξη. Ας κάνουμε λοιπόν κοινή συζήτηση για τα τρία θέματα που αφορούν την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Θα καλέσω την κυρία Μπιλμπά, τον κύριο Ρικέ και την κυρία Γιούτο, τους ηγητές, να παρουσιάσουν τα κείμενά τους. Μετά θα δώσω το λόγο στους διάφορους σκιώδεις ηγητές κατά σειράν πολιτικών ομάδων και στους άλλους βουλευτές που τα επιθυμούν που θα λάβουν το λόγο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμών για την παρουσία του. Πού είναι? Ευχαριστώ. κυρία μου, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είστε για την ΕΟΚΕ θα μας κάνετε μια σύντομη παρέμβαση τρίλεπτη. Σύντομη και περιεκτική. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Θα έχετε στη διάθεσή σας περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση. Δίνω το λόγο στις συζητητές. Ξεκινούμε με εσά, κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό απόγευμα και βεβαίως να συλληπιθώ κι εγώ με την ίδια αλληλεγγύη που το έκανε η Πρόεδρό μας. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, αυτή η οδηγία είναι μία αναθεώρηση ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων σύμφωνα με το REFIT το οποίο έχει ως σκοπό να κωδικοποιήσει, απλουστεύσει και βελτιώσει την νομοθεσία μας. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν είμαστε κι εμείς σύμφωνοι. Εμείς προκρίναμε πολλές από αυτές τις αλλαγές στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας και ε, επειδή έχουμε ασχοληθεί με τα διάφορα πακέτα για την ασφάλεια, ζητήσαμε να έχουμε και μια νομοθετική ε, πρόταση έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε στις νέες αυτές ε, διατάξεις τις ε, σχετικές για την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατικά πλοία. Έχουμε λοιπόν την ψηφιακή καταγραφή που είναι μια νέα διαδικασία μέσω μιας εναρμονισμένης διαδικασίας με την ενιαία εθνική θηρίδα και πρέπει να σας πω πως το σύστημα που ε, καταχώρησης που έχουμε αυτή τη στιγμή και καταγραφής ατόμων από τις εταιρείες θα αντικατασταθεί από μια καταγραφή σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μεταδίδεται στους, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στις αρμόδιες αρχές όταν το επιθυμούν από την ε, ενιαία εθνική θηρίδα. Η πρόταση την οποία ε, συζητάμε είναι μια πρόταση η οποία σε πολλά σημεία μας βρίσκει σύμφωνους ε, για τις διατυπώσεις υποβολής, για παράδειγμα, και για το πεδίο εφαρμογής που προτείνεται. Τώρα, να σας πω καταρχήν πως ε, συμφωνούμε και με την πρόθεση της επικαιροποίηση, της ενημέρωσης και της απλούστευσης σε όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα. Θεωρούμε πως με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, η τεχνολογική κοινοτομία θα πρέπει να αποτελέσει κομβικό σημείο αυτή τη έκθεση, γιατί όλοι έχουμε δει πόσο σημαντική είναι Μιλάμε για την περίπτωση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, των διαφόρων ρομπότ, τα drones, τα οποία έχουμε ε, πια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτάσεις που κάνουμε και μιλάμε και για την ψηφιακή καταγραφή μέσω της Εθνικής Ενιαίας ε, Θηρίδας, όταν ξεπερνά ο πλούς τα 20 μίλια. Επίσης θα πρέπει εμείς να στοιχηματίσουμε υπέρ αυτών των αλλαγών σε εθνικό επίπεδο μέσω μιας πλατφόρμας η οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί ε, με τον ίδιο τρόπο, αλλά όχι πλέον μέσω ευρωπαϊκή, ε, εθνικής ε, μέσω μιας ευρωπαϊκής ενιαίας Γιατί νομίζω ότι αυτό αποτελεί τη λύση για το μέλλον και το έχουμε δει και με άλλες αντίστοιχε εκθέσεις. Εν πάση θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο να είμαστε πιο ευέλικτοι για τους ε, μεταφορείς, για παράδειγμα, για πιο ε, σύντομα ταξίδια και έχουμε και μια τρίτη εναλλακτική λύση γιατί μιλήσαμε και με τους εμπλεκόμενους που επηρεάζονται από την πρωτοβουλία αυτή. Μια τρίτη λοιπόν εναλλακτική λύση έτσι ώστε να έχουμε δηλώσεις ε, μέσω των συστημάτων των ηλεκτρονικών που έχουν εγκριθεί ήδη για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα εφιστάμενα συστήματα διατύπωσης και υποβολής δηλώσεων αρκεί να έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά και ταχύτατα έτσι ώστε να μην ε, παραλύσει αυτή τη στιγμή η βιομηχανία, αλλά θα πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι αποδεδειγμένα ασφαλή και σίγουρα, γιατί μιλάμε εδώ για περίπτωση τοπικών δρομολογίων που δεν επηρεάζουν την ευρύτερη ε, τις ευρύτερες μεταφορές της ε, περιοχής. Τώρα, για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ε, στα πλαίσια των στόχων αυτής της οδηγίας και θα πρέπει αυτομάτως να διαγράφονται όταν δεν χρειάζονται πια για το σκόπο για, το σκοπό για τον οποίο έχουν καταγραφεί. Επίσης, οι πληροφορίες που στέλνονται για άτομα ή πολίτες που έχουν ανάγκη συγκεκριμένης βοήθειας και για κάποιες επίγουσες καταστάσεις να σας πω πως τις οδηγίες, στην οδηγία αυτή τη στιγμή λένε πως τα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες θα πρέπει με εθελοντικό τρόπο να καταθέτουν τις πληροφορίες αυτές προς καταγραφή. Να σας πω πως από τη στιγμή που έχουμε κάποιο είδους ατύχημα ή συμβάν ε, ή κάποιο επεισόδιο και τα άτομα αυτά χρειάζονται ειδική βοήθεια και αυτό δεν έχει προβλεθεί, τότε και η δική του ασφάλεια διακυβεύεται και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να, ληφ, να ληφθεί δεόντω υπόψη και να του βοηθάμε με τον ίδιο τρόπο που βοηθάμε του υπόλοιπου. Ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται, είναι δύσκολο να γίνει δεκτό και είναι ε, ένα σημείο ε, αμφισβητή ζητούμενο, αλλά νομίζω πως θα πρέπει και εδώ να φανούμε αρκετά αυστηροί. Επίσης, για τη διάρκεια πέντε χρόνια, το οποίο θα, πέντε χρόνια διάρκεια που θα μπορεί να παραταχθεί ε, βεβαίως μετά από έγκριση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρει μήνε θα είναι ο χρόνο που θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διάθεσή τη ε, για τι ε, προτάσει των κρατών μελών και για τι κυρώσει που ενδεχομένω θα επιβληθούν ή για περίπτωση στρέβλου ανταγωνισμού. Νομίζω ότι μια μεγαλύτερη διάρκεια μπορεί ε, να είναι προβληματική και τέλο. η για περιπτωση στρεβλου ανταγωνισμου νομιζω οτι μια μεγαλυτερη διαρκεια μπορει να ειναι προβληματικη και τελο η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας και θα καταθέσει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο σε δύο χρόνια από τη στιγμή της εφαρμογής. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μία μείωση της προθεσμίας και όχι μετά από τα 7 χρόνια τα οποία αυτή τη στιγμή έχει συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία τούτου της πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπιλμπάου. Τώρα η κυρία Γιούτο για τους κανόνες προδιαγραφής ασφαλείας για την επιβατικά πλοία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη ε, κάνει μία πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών και εκεί είχαμε την ε, δυνατότητα να εξετάσουμε από κοινού την κατάσταση. Ε, τώρα λοιπόν επανεξετάζουμε την οδηγία 45 η οποία ορίζει τις προδιαγραφές ε, ασφάλειας ε, για τα επιβατικά πλοία τα οποία έχουν κατασκευαστεί από χάλιβα ή από παρεμφερές υλικό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να προβλέψει κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή ε, τι δεν προβλέπει αυτή η οδηγία. Η πρώτη εξαίρεση αφορά όλες, όλα τα σκάφη ε, τα οποία είναι πάνω από 18 περίπου μέτρα. Και επειδή αυτό είναι ε, τεχνικό επίπεδο, όσα είναι λιγότερα από 24 μέτρα δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές όπως τα μεγαλύτερα σκάφη. Η δεύτερη εξαίρεση αφορά τις τα σκάφη εκείνα τα οποία μεταφέρουν προσωπικό σε εργασία, στο χώρο εργασία και αυτοί δεν είναι οι κανονικοί επιβάτε, είναι ειδικό προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση που δεν ορίζεται επακριβώ, τουλάχιστον όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των εργαζομένων. Ω εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει αυτού να του εξαιρέσει. Τώρα, όσον αφορά τι άλλε εξαιρέσει, υπάρχει πρόταση να αποκλειστούν και τα τέντερ, τα μικρά τα σκαφάκια τα οποία μεταφέρουν τα, ε, το επιβατικό προσωπικό από τα μεγάλα σκάφη ε, στα κουρασγερόπλαια στις ακτές. Μετά τα ιστιοφόρα, ε, τα οποία και αυτά έχουν κάποιες ειδικέ προδιαγραφές και εκεί πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια γιατί υπάρχουν κάποιες ε, γκρίζες ε, φές ζώνες οι οποίες ε, είναι κάπως προβληματικές. Υπάρχουν πολλές εμφωλίες από αυτόν τώρα. Όσον αφορά αυτά που περιλαμβάνονται, θέλουν να περιλαμβάνουν εκείνα τα σκάφη που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, γιατί αυτό θεωρείται ότι είναι ισοδύναμο του χάλιβα. Και τέλος υπάρχουν τα ε, σκάφη ανοιχτή θάλασσα. Αυτή είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όσον αφορά τη δική μα την πρόταση, υπάρχουν τρία θέματα που εστιάζουμε την προσοχή μα. Το πρώτο είναι ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν προδιαγραφέ για τι ε, εξαιρέσει. Δηλαδή να μην αφήσουμε κενά, να είμαστε σίγουροι και να ξέρουμε ότι εδώ πρόκειται για διεθνεί προδιαγραφέ. Άρα δηλαδή αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν σημεία αναφορά και προδιαγραφέ ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσφέρει την κατευθυντήρια γραμμή και τις προδιαγραφές ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, δηλαδή να μην αφήσουν γκρίζες ζώνες. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στη διαφάνεια. Για να υπάρχει μέγιστη δυνατή διαφάνεια, οποιαδήποτε εξαίρεση ή οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται θα πρέπει να δημοσιεύεται σε, ε, στο διαδίκτυο. Και τέλος, όσον αφορά τον κοινωνικό χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει προορατικά ε, θα πρέπει να προάγει τις σωστές συνθήκες εργασίας, τη σωστή ενημέρωση. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες και το προσωπικό θα μπορούν να ε, ταξιδεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτό βέβαια δεν είναι δεδομένο γιατί ξέρουμε ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πέρα από την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει και μια σαπή θέση του Συμβουλίου η οποία αναφέρεται σε ε, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο ζητάει δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη αφορά το αλουμίνιο που θεωρείται ισοδύναμο υλικό. Επ' αυτού η Γαλλία ζητάει μία εξαίρεση για 14 χρόνια για να μπορεί να προσαρμοστεί, να κατασκευάζει τα σκάφη από αλουμίνιο. Και η δεύτερη εξαίρεση αφορά ε, τον θαλάσσιο χώρο. Εκεί γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας. Δηλαδή η γεωγραφική θέση της Ελλάδας με όλα αυτά τα νησιά που έχει ε, δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν όλες αυτές οι διατάξεις. Και γι' αυτό λοιπόν ε, έχει προ προταθεί να υπάρξουν ειδικοί ορισμοί για την ε, Ελλάδα. Τώρα για τα άλλα κράτη-μέλη υπάρχει σαφώς οριζόμενος θαλάσσιος χώρος. Και όσον αφορά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όπως σας είπα, υπάρχουν σαφείς ορισμοί και τόσο στην πρόταση του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνονται άλλα ε, διαφορετικά στοιχεία. Αυτά σε γενικές γραμμές προς τα εκεί κατευθυνόμετα. Όπως σας είπα υπήρξε ήδη μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών. Ε, δεν μπορούσαμε να τοποθετηθούν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούτο. Ο κύριος Ρικέ τώρα είναι εισηγητής μας για το σύστημα επιθορήσεων για την των τακτικών δρομολογίων διασυνοριακών συγκοινωνιών και χρήση σκαφών υψηλής ταχύτητας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να επενθυμίσω τον όλο ιδιαίτερο χαρακτήρα των, αρμα... των αχηματαγωγών και που δημιουργούν ειδικού κινδύνους Πολλά ατυχήματα είχαμε πολύ θεαματικά στην Ευρώπη όσον αφορά αυτά τα σκάφη τα τελευταία χρόνια και κάθε φορά τα θύματα είναι εκατοντάδε. Άρα είναι ένα ιδιαίτερο θέμα να επενθυμίσουμε ότι τα ρορό επίσης είναι σκάφη που μεταφέρουν και επιβάτες διότι μεταφέρουν και τους οδηγούς των φορτηγών. Οπότε μπορούμε να έχουμε 200 με 300 οδηγούς ε, ε, φορτηγών. Οπότε γίνεται το οχηματαγωγό και επιβατικό πλοίο. Λοιπόν, θέλουμε καλύτερη νομοθεσία και καλύτερη ρύθμιση και θέλουμε να διατυπώσουμε τις προηγούμενες οδηγίες που είχαν αφήσει να συνεπάρχουν οι οδηγίε και δημιουργούσαν νομικές, ε, και, ε, νομικά κενά και επικαλύψεις. Προτείνει να καταργηθεί η 1999-35 που προβλέπει ειδικές, περιφ... ρυθμίσεις για τη και τα ταχαία σκάφη και το 2016 όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου να επιβάλλονται τα μέτρα. Υποστηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει στο στόχο την εξασφάλιση κοινών σαφών απλουστευμένων ενισχυμένων κανόνων χωρίς να υπάρχουν νομικά κενά αλλά χωρίς να δημιουργούνται και πλεονασμοί. Λοιπόν, κάποιες διευκρινήσεις θέλαμε να κάνουμε όσον αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν σαν στόχο τη διευκρινήση του κειμένου κυρίως όσον αφορά τον ορισμό των αρμοδίων αρχών ε, και το κόστο το ενδεχόμενο για τους λιμένες ε, και κάποια κείμενα που ίσως να αφήνουν αφησιμίες και να οδηγούν σε σύγχυση. Λοιπόν, ε, ποια είναι τα θέματα τα βασικά που πρέπει να εξεταστούν. Το άρθρο 5 της παραγράφου 1 που καλύπτει αβεβαιότητα και κενά λέει ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δύο επιθεωρήσεων ούτω ώστε να μην γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο επιθεώρηση. Δεν έχει νόημα. Ανα... Υπάρχει επαρκέ περιθώριο λιγμών, ούτω ώστε μεταξύ των δύο επιθεωρήσεων υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, ούτω ώστε πράγματι να γίνονται τα δέοντα. Πρέπει να γίνεται κάθε εξάμεινο δύο έλεγχοι το χρόνο με ένα περιθώριο ε, λιγμών ενό μήνα. Δηλαδή μπορεί να γίνεται κάθε πέντε μήνε, εφτά μήνε, να περάσουν πέντε μήνε, εφτά μήνε μεταξύ των ελέγχων είναι το πρόβλημα ε, προβλήματα όσον αφορά τη χρήση αυτών των πλοίων ε, της περίοδου υψηλής κινδύνου. Οπότε πρέπει αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη στη συχνότητα των ελέγχων για να μην δημιουργούμε στους πλειοκτήτες και στους ναυλωτές προβλήματα. Να έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια για να λάβουν υπόψη ε, και τις ανάγκες συμπορικές και να έχουν και περιθώριο ώστε να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα δύο. Το άρθρο 5 της παραγράφου 3 μετά υπάρχει απαλλαγή από τον έλεγχο όταν αλλάζει ο προορισμό του σκάφους. Και αυτή δεν θα πρέπει να χορηγείται διότι οδηγείται έτσι έχουμε ανήσει μεταχείριση κάποιων κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια κάτι μέλη που θέλουν να επανελέγχουν το σκάφος ούτως ώστε να γνωρίζουν ότι το σκάφο αυτό ε, συμφωνεί ε, με τους προδιαγραφές ασφαλείας. Κλείνοντας, Έχα κάνει διάφορα, λοιπόν, στα λιμάνια για επιθυρώσει και κατά διακάτης υπηρεσία. Έχω συμμετάσχει αυτά και μου έχουν εξηγήσει και οι κυβερνήτες και τα πληρώματα ελέγχου τα προβλήματα. Είπαμε να υπάρχει και ένα περιθώριο αυτό που είπαμε των δύο μηνών, συνυπλήν, και κάτι πιο περίπλοκο, ότι δίνει ποσοστώσεις για ελέγχου στα κράτη-μέλη, αναλογικά με τον αριθμό των σκαφών που είναι σε υπηρεσία στο συγκεκριμένο λιμάνι κράτους μέλους και η Ένωση εξακριβώνει τα κάτι μέλη καλύπτουν τις ποσοστώσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτές οι ποσοστώσεις βασίζονται σε προτεραιότητες 1 και 2 που εμπεριέχουν αυτές οι προτεραιότητες. Είδη σκαφών και συχνότητα ελέγχων. Και αντιλαμβανόμεθα ότι τα σκάφη, τα επιβατηγά που συζητήσαμε που έχουν ιδιαιτερότητα στον αφορά ασφάλεια δεν θεωρούνται συστηματικά σαν σκάφη με υψηλό κίνδυνο στον αφορά την ασφάλεια. Ενώ αυτό ισχύει. Άρα τα κράτη-μέλη πολύ συχνά έχουν την επιλογή μεταξύ ε, δύο ελέγχου μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο να ελέγχουν τα σκάφη, κάτι που είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν, εάν θέλουν να συμπληρώσουν την ποσόστοση, να μην γίνεται ο έλεγχο ετησίω. Θέλουμε λοιπόν στην οδηγία να εισάγεται μια δυνατότητα αυτά τα σκάφη που έχουν, αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερους κινδύνου να μπουν στην κατηγορία 1 κατηγορία ψηλού κινδύνου, ούτω ώστε να μπαίνουν στην ποσόστοση με προτεραιότητα. Γιατί, διότι τα κάτι μελη τώρα αντιμετωπίζουν πολύ συχνά επιλογή, δίλημα, ή να μην ελέγχουν όλα τα, τα οχηματαγωγό, ε, ή δεν συμπληρώνουν τι ποσοστώσει γιατί μόνο τα οχηματαγωγά και τα ferry ελέγχουν και δημιουργούνται προβλήματα στου σωστού στι 1 και 2. Είναι περίπλοκο, το παραδέχομαι, αλλά η κεντρική ιδέα είναι να θεωρήσουμε ότι τα σκάφη θα πρέπει να έχουν προτεραιότητε ελέγχου λόγω εξαιρετικά υψηλού κινδύνου που θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί. Διότι αν δεν ελέγχονται τακτικά αυτά τα σκάφη, αντιπροσωπεύουν πολύ ε, ψηλό κίνδυνο. Είχαμε συναντήσει με του κοιόδη, θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα τη προσέγγιση. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα, αυτό ο κανονισμό. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ερικέ. Θα αρχίσει λοιπόν η συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με εσά, κύριε Μπόγκλης. Μη διστάζετε, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι εδώ για να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σχετικά με την πρόταση τροποποίηση οδηγία 45 του 2009. Πιστεύω ότι είναι μια πρόταση που στο σύνολό της μπορεί να υποστηριχθεί, διότι επιτρέπει να εξαλείψουμε κάποιες αμφισημίες που υπήρχαν ε, στο αρχικό κείμενο της οδηγίας, που οδήγησαν σε ερμηνείες ποικίλε από πλευρά των διαφόρων εθνικών αρχών αν θέλουμε το βασικό στόχο, την προτεραιότητα, δηλαδή να αγγιθούμε υψηλό επίπεδο ασφαλεία για του επιβάτε και το προσωπικό, θέλουμε αυτό. Ταυτόχρονα όμω θέλουμε και μια πλούστευση και μια μείωση τη γραφειοκρατία όσον αφορά το ολοπλαίσιο και μειώνοντα και το συμπληρωματικό κόστο. Οπότε συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά την πρόταση να εξαιρέσουμε τα επιβατικά σκάφη με μήκο μικρότερο από 24 μέτρα. Συμφωνώ με την εξαίρεση των offshore, των οχημάτων και τα μικρά σκάφη ίδια που εξυπηρετούν τα κρουαζιερόπλια και ε, συμφωνώ με την αντίληψη που παρουσιάστηκε για το πεδίο εφαρμογή του αποβράσου του κειμένου για τα σκάφη από αλουμίνιο. Εγώ συζήτησα με την εισηγήτρια, διάβασα τις προτάσεις της, για τροπολογίε που ε, διατυπώθηκαν και μπορώ να τα υποστηρίξω αυτά κυρίως όσον ακολουθούν την κατεύθυνση εγγύησης μεγαλύτερης διαφανείας και πάνω απ' όλα καλύπτεται η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει προσανατολισμού στα κράτη-μέλη προ εναρμόνιση των διατάξεων, κυρίω όσον αφορά τα σκάφη που είναι μικρότερα από 24 μέτρα. Βεβαίω θα συζητήσουμε και τι άλλε τροπολογίε που θα υποβληθούμε στις 9 Μαρτίου, αλλά στο σύνολό τη η πρόταση αυτή μπορεί να τύχει υποστήριξη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο. Στην κυρία Μοντέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Δεν ξέρω αν έχω δύο λεπτά χρόνο στην διάθεσή μου, γιατί η παρέμβαση που θα κάνω είναι διπλή. Δηλαδή, θα ήθελα να μιλήσω και για τα όσα είπε η κυρία ε, Μπιλμπάου και όσα είπε ο κύριος Ρικέρο. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θα τα σχολιάσω και τα δύο ταυτόχρονα. Λοιπόν, να σας πω πως καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφη την κυρία Μπιλμπάου για την παρουσίαση που έκανε του θέματος και νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου. Να σας υπενθυμίσω δε τα εξής. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, πως ε, δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην κυκλοφορία ε, σκαφών μεταξύ νησιών για παράδειγμα ή για κάποια πολύ σύντομα ταξίδια. Και το γεγονός πως θα πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία πριν τον απόπλου των σκαφών νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται μέχρι 10 λεπτά πριν τον απόπλου. Είναι σωστό αυτό να το λάβουμε υπόψη, γιατί τι γίνεται με τα κρουαζιερόπλια για παράδειγμα. γιατί νομίζω ότι για το κροζιερόπλαιο πιο συγκεκριμένα αυτή η διάταξη είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Τώρα, ε, και... Έχουμε ήδη ζητήσει τη γνωμοδότηση του IMO για να δούμε για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε μέχρι και την ε, ημερομηνία γέννησης και όχι μόνο την υπηκότητα. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να λέμε μόνο το έτος γέννησης, είναι ανάγκη να δίνουμε ολόκληρη την ημερομηνία. Και έχω και άλλη μια ερώτηση ε, για τα 20 μίλια και νομίζω αυτή θα πρέπει να την ε, απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέει ο ΑΕΜΟ? 20 μίλια από την ακτή. Αυτός δεν είναι ο διεθνής κανόνας. Γιατί δημιουργούμε εμείς ένα νέο κανόνα εμείς στο κείμενό μας. Και τέλος, για τα όσα μας είπε ο κύριος Σερκέρ. Μιλήσατε για σηματαγωγά ρορό και για τα χύπλοα. Κοιτάξτε, σε συγκεκριμένες εποχές δεν ξέρω εάν είναι δυνατόν να δώσουμε κάποιες εξαιρέσεις μέσω της οδηγία μας ή αν θα έπρεπε οι επιθεωρήσεις να γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί όπως σας είπα είναι εποχιακά δρομολόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχήν που με προειδοποιήσατε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Η κυρία Αγέντε είναι η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα να σας πω πως για την έκθεση της κυρίας Αγιούτο θα ήθελα απλώς να την ευχαριστήσω γιατί έχει κάνει κάποιες προτάσεις και να σας πω πως το μόνο που με ανησυχεί είναι Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μέσω του Refit προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευκρίνεια, αλλά εδώ έχουμε πολλούς αποκλεισμούς από το πεδίο εφαρμογή οδηγία και αυτό το στοιχείο μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο ασφάλειας εάν δεν, ε, κάνοντας παράλληλα τέτοιου είδους εξαιρέσεις. Είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά πολύ συχνά ε, οι κανόνες ε, ε, για την εξασφάλιση ενός καλού επίπεδου ασφάλισης μας οδηγούσαν, μας οδηγούσαν στο να εισάγουμε κάποιες αρκετά αυστηρές διατάξεις και δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί έχουμε τόσες πολλές εξαιρέσεις από την οδηγία. Και βέβαια θα στηρίξουμε την κυρία Αγιούτο. Ναι, σίγουρα χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα βοηθήσουν στο να εναρμονίσουμε ε, για παράδειγμα το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας ε, για τα σκάφη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή. Επίσης, θέλω να επαναλάβω πω υπάρχει μια ανάγκη και στον IMO για αυτά τα ε, σκάφη τα οποία ε, ουσιαστικά τι κάνουν ε, στην ανοιχτή θάλασσα ανεφοδιασμό να συμπεριλάβουμε κάποιους κανόνες έτσι ώστε και εδώ να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας γιατί σίγουρα οι κίνδυνοι είναι πολλοί γιατί βεβαίω, επειδή όλα αυτά είναι στην ανοιχτή θάλασσα ή offshore, ε, καταλαβαίνετε ότι εκθετικά ανεβαίνει ο κίνδυνος και έχουμε σκάφη τα οποία μεταφέρουν για παράδειγμα προσωπικό ε, που αποτελούν ένα φαινόμενο όλο και πιο συχνό. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και εδώ να προτείνουμε κάτι για να συμπεριληφθούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Επίσης, ε, για τα σκάφη από αλουμίνιο. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, εδώ είμαστε στα πλαίσια του refit της νομοθεσίας, αλλά έχουμε τεχνικές μελέτες για τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ασφάλεια ε, για τα σκάφη με κήτος από χάλιβα ή με κήτος από αλουμίνιο έτσι ώστε να γνωρίσουμε ποια θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ στην οδηγία γιατί για το κήτος που είναι από αλουμίνιο για παράδειγμα για σκάφη αλίας εκεί είχαμε μια αύξηση του αριθμού ατυχημάτων και θα ήθελα να δω αν έχει γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό κάποιος ή αν το έχει μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Σαϊόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μιλήσαμε, συνομιλήσαμε με τους συναδέλφους, έγιναν διάφορες επαφές με τους ενδιαφερομένους, οπότε επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις ε, απόψεις τους. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση της κυρίας ε, Μπιλμπάου είναι πολύ καλή. Αναφέρεται σε όλα τα ενδιαφέροντα ζητήματα. Δεν θα πω με ποια σημεία συμφωνώ, με ποια διαφωνώ, δεν έχουν πολύ χρόνο. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που εκεί θα πρέπει το κείμενο να γίνει πιο σαφές. Για την ενιαία θηρίδα, ευρωπαϊκή ενιαία θηρίδα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το σύστημα, να μιλήσουμε και για τα εθνικά συστήματα για ενιαία θηρίδα. Πώς λοιπόν το, ε, το κρατικό, το εθνικό ε, σύστημα ενιαίας θηρίδας θα γίνει ευρωπαϊκό, Ποια θα είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ενιαία στηρίδας. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε πολλά συστήματα για φύλαξη στοιχείων και θα ήθελα να γνωρίζω τι γίνονται αυτά τα στοιχεία, αυτά τα δεδομένα και τι πρέπει να γίνεται μετά από χρονικό διάστημα με αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να διαγράφονται τα δεδομένα μετά κάποια χρονική περίοδο. Πώς και μετά ποια χρονική περίοδο. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Βλέποντας τώρα τις προθεσμίες, έχουν βραχυνθεί όλες. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, συμφωνούμε, αλλά αν παραμένει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία των δεδομένων. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει την άποψή της. Συμφωνεί με αυτή τη βράχυνση, τον περιορισμό των χρονικών ορίων. Ιδού λοιπόν Αυτά ήταν ε, όσα είχα να πω στα πρώτα μου δύο λεπτά. Και μετά στο, πάω στον κύριο Ρικέ. Νομίζω έχω άλλα δύο λεπτά για τον κύριο Ρικέ. Διότι είμαι ακόμα σκιώδη ηγητή των σοσιαλιστών. Έχετε δύο λεπτά παρέμβαση. Δεν είναι δύο λεπτά ανά παρέμβαση. Συμφωνείτε. Δύο λεπτά στη γενική σας παρέμβαση. Κύριε Βιχεβή, όλοι ξεπέρασαν τον χρόνο τους και δεν θέλω να το ξαναφέρω το θέμα. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να θέσετε το ερώτημά σας προς τον κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ όμω ότι αυτό είναι πολύ άδικο. Θα ήθελα να έχω δύο φορέ δίλεπτο, διότι είμαι σκιώδη ηγητή για δύο θέματα. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα, τι να πω, να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για το έργο που έκανε, που σωστά αναφέρεται στον παράλληλο χαρακτήρα των δύο κειμένων. Συμφωνούμε λοιπόν με την άποψη του κυρίου Ρίκε. Δεν χρειαστήκατε καν το δίλεπτο για να πενέστε το έργο του κυρίου Ρικέ. Η κυρία Φώστερ, εσείς έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Η κυρία το Μπίκ θα συντάξει την πρώτη έκθεση και εγώ τελευταία και εκείνη θα πάει στην Επιτροπή Ελίες. Είναι εκείνη η ε, πρώτη γιατί Είναι η σειρά τη να μιλήσει. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου και θα μιλήσω μόνο για αυτή την έκθεση. Χαιρετίζω λοιπόν τον ε, στόχο αυτή τη οδηγία, που είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών ε, και να μην βρίσκεται σε κίνδυνο η ασφάλειά του λόγω υπερβολικού ε, βάρου και σε περίπτωση ατυχήματο να υπάρχουν και απαραίτητε ενέργειε. Θα πρέπει λοιπόν οι πληροφορίε να δίδονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων υπό τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο στόχο είναι να είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίε σε περίπτωση ατυχήματο χαιρετίζω την έκθεση ε, ξεκάθαρη κανόνες, ε, κυρίως ε, όσον αφορά και την διατήρηση των στοιχείων των επιβατών και από την Ατυλική Εταιρεία και από τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύονται τα μικρά σκάφη από την αυξημένη γραφειοκρατία και να χαιρετίζουμε τις εναλλακτικέ λύσεις. Οι πληροφορίες για τα άτομα που επιβαίνουν στο πλοίο θα πρέπει να προστατεύονται από τελειοφθορά και από την πειρατεία. Πολύ ωραία. Ε, κύριε Φώστερ, εγώ ε, ε, θα απαντήσω στον κύριο Ρικέ μεταξύ ε, άλλων. Όσον αφορά τα ρόρο, θέλω να σας πω ότι είναι πια πάρα πολύ καλή έκθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία από αυτού και σε γενικέ γραμμέ ε, όλα αυτά θα τα στηρίξουμε. Όσον αφορά την κυρία Τότο, νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή ε, συζήτηση για, ανάμεσα στου Κιώδη. Έδειξε πάρα πολλά θέματα η ίδια, ε, θέματα ασφάλεια και χαιρετίζουμε τη θέση του Συμβουλίου και τη Κομισιόν σχετικά με το να αλλάξουν κάποιε κατεξοδότηση πράξει σε πράξει εφαρμογή, εφαρμοστικέ πράξει. Επίση, χαιρετίζουμε και εμεί αυτές τις ε, αλλαγές. Όσον αφορά τώρα τις προδιαγραφές, το να υπάρχει επιπρόσθετο, πρόσθετο εξοπλισμός ασφάλειας, αυτό εξαρτάται και από το ύψος και έτσι φτάνω τώρα στις εξαιρέσεις. Πολύ σωστά λοιπόν έγινε λόγος για τις εξαιρέσεις, το κατά πόσον θα εξετάζουμε τα μικρά σκαπάκια αυτά, τα τέντερ ή τα ιστιοπλώα. Ε, ιστιοπλοϊκά. Νομίζω ότι εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει συμμόρφωση με τους ε, προδιαγραφούς του IMO. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταλήξουμε τελικά σε μια περιγραφική κατάσταση όπου δεν θα συμμορφωνόμαστε με τις κανόνες ε, του IMO. Έχουμε σαν παράδειγμα τα κλασικά σκάφη. Και όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διαφάνεια, αλλά εξαρτάται βέβαια από το ποιο ε, θα μπορεί να παίρνει αυτέ τι ε, πληροφορίε. Γιατί υπάρχουν και θέματα ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι όλοι μπορούν ε, να μπαίνουν στο διαδίκτυο και να αποκτούν αυτέ τι πληροφορίε. Δεν είναι σωστό αυτό. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το, την σκιώδη συγγήτρια. Τα συζητήσαμε τα θέματα εκτενώ και θα δούμε πώ θα προχωρήσουμε συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοινώνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές και να σας πω πως ε, κυρίως τα έγγραφα αυτά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι ένα θέμα το οποίο καλώς κάνει και μας απασχολεί γιατί εμείς πρέπει στο επίπεδο της ασφάλειας να κάνουμε κάθε προσπάθεια να βελτιώσουμε τα επίπεδα ασφάλειας όχι μόνο ε, των επιβατών αλλά και των πληρωμάτων. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εκείνες τις βελτιώσεις που χρειάζεται το κείμενο. Ε, μιλώ για το Μητρό γιατί βέβαια υπάρχει η υποχρέωση καταγραφής των επιβατών και νομίζω το σημείο αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες ισορροπίες έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε υπερβολικό διοικητικό βάρος στους ε, ε, επιχειρηματίες και στους ε, πλειοκτήτες στα κράτη-μέλη. Για να εξοικονομήσω δε κάποιο χρόνο, νομίζω ότι Μπορώ να σας διαβάσω και τα όσα μας έστειλε ο κύριος Στελίου στα αγγλικά, ο οποίος ευχαριστεί πολύ για τα όσα έκαναν οι συγητές. Ο κύριος Ρικέ έχει μια ερώτηση. Θέλω ένα καφέ να μου να με κεράσει κυρία Αγιούτο γιατί πρέπει να σας πω πως ε, Πρέπει να σας πω πως αν εξαιρέσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία τα οποία θα ήθελε να εξαιρέσουμε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμπεριλάβουμε το αλουμίνιο και το λέω, θα σας το πω γιατί γιατί είναι κάτι το οποίο θα ανησυχήσει όλα τα ναυπηγεία στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν αλουμίνιο στην κατασκευή πλοίων κυρίως βέβαια τα γαλλικά ναυπηγεία εντάξει ας είμαι ειλικρινή στο σημείο αυτό οπότε νομίζω πως το σημείο αυτό το κατά πόσο θα συμπεριληφθεί το υλικό αυτό ή όχι έτσι μόνο του πρέπει να κάνουμε παραπάνω συζήτηση. Γιατί δηλαδή όχι κάποια άλλα υλικά. Ε, δεν νομίζω ότι το να, στο να ακολουθήσουμε ό,τι κάνουμε με το χάλιβα είναι σωστό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιου αποκλεισμού. Αν το κάνουμε θα μπορούσαμε πάντως να δώσουμε μια συγκεκριμένη ε, προθεσμία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο αντικειμενικοί μέσα στην υποκειμενικότητά μα. Uh, thank you, Chair. Um, yes, well, θα αναφερθώ και στις τρεις οδηγίες ε, για το, και το Refit. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να υποβάλω και δύο θέματα γενικής φύσεως. Πρώτα απ' όλα, παρότι αναγνωρίζω ότι η εκπαίδευση προσωπικού για να μπορέσουν να είναι ικανά σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος ασφάλειας, αυτό δεν εμπίπτει βέβαια στις, ε, σε αυτή την Αλλά εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΜΣΑ οφείλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την εκπαίδευση των ατόμων και την κοινωνική τους κατάσταση που απασχολεί σε αυτόν τον τομέα. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι πολύ σωστά εκπαιδευμένο για να ε, βοηθάει αποτελεσματικά τους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βελτιωθεί ο ε, υπερεθνικός συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες παροχής ε, βοήθειας γιατί και τα ποτάμια και οι θάλασσες και αυτά παίζουν ρόλο σε θέματα ασφάλειας, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ε, ασφάλεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζει ασφάλεια και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις μου, κατανοώ βέβαια πολύ καλά ότι η πρόθεση του REFIT είναι να απλουστευτεί η κείμενη νομοθεσία και αυτή να ε, προσαρμοστεί και στους κανόνες του ΑΕΜΟ. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον και πώς ε, αυτό όλο, αυτές οι τροπολογίες θα βελτιώσουν την εφαρμογή των ε, οδηγιών. Αυτή είναι κυρίως μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Και τέλος, ε, θα ήθελα να γνωρίζω ε, κατά πόσον θα αποφασίσουμε ως Επιτροπή αν είμαστε υπέρ των κατεξουσιοδότηση ή των εφαρμοστικών πράξεων. Αυτά είχα να ρωτήσω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Η κυρία Γνωτού. Ευχαριστώ τειλορ η κυρια γνουτου Πρόεδρε. Οι δύο οδηγίε που τροποποιούνται καθώς και νέα οδηγία όσον αφορά τους ελέγχους για θέματα ασφαλείας εν γέννη επιτυχαίνουν τους στόχους τους. Οι προτάσει των τριών εισηγητών θεωρώ ότι είναι κάτι αναγκαίο και σχετικό. Όσον αφορά την καταχώρηση των επιβατών, την επιθυμία της κ. Μπιλμπάου για τρίτο τρόπο διαβίβασης στοιχείων των ταξιδιωτών, καθώς και την εξασφάλιση καταστροφής αυτομάτου και ταχείας των δεδομένων, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και θα διευκόλυνε την πραγματική εφαρμογή της οδηγία όσον αφορά τους ελέγχους περιασφαλείας, ο συνδυασμό των ελέγχων ε, έχει ήδη περιορίζει τους χρήστες και, και οι προθεσμίες για την κατασκευή πράξης που προτείνονται από, από τον κύριο Ρικέ επιτρέπουν καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο παρόλο που αυτό παραμένει θεωρητικό λόγω τεχνικού χαρακτήρα του τομέα που προσπαθούμε να καλύψουμε. Ανησυχώ λίγο για την πρότασή σας διαχωρισμού του, ε, του ελέγχου και του χρήστου του πλοίου και του ναυλωτού. Ε, δίνεται μεγάλη ευελιξία εκεί, αλλά ίσως ε, εάν υποχρεωθούν οι ναυλωτές να πηγαίνουν σε πιο φιλικό λιμάνι και να οδηγούνται σε χρήση ε, κρυφών επιδοτήσεων, όπως γίνεται με τις εταιρείες low μετά έχουμε την πρώτη κυρία Σαγιούτο που δίνει θετικά στοιχεία στον αυτά τα θέματα ασφαλείας σε μια οδηγία η οποία ήδη είναι καλή. Αντίθετα, η συμπεριλήψη των σκαφών από αλουμίνιο εντός της οδηγίας θεωρώ ότι θα ήταν κάτι επιβλαβές οικονομικά και δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί εκτός από το τίμημα που αναφέρατε ε, κύριε ε, Ρικέ θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίες και το ίδιο για τα σκάφη λιγότερα, τα μικρότερα από 24 μέτρα εξαίρεση αυτών ε, θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Και έτσι άλλες δύο οδηγίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη διάρκεια των κατεξιζώτης συμπράξεων και να προωθήσουμε την πρώτη αξιοδότηση που καθορίζεται στην επταετία. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ απόμακρο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κύριε Ντεμόντε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές ε, και τους και οδησηγητές. Δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Μία αφορά και τις τρεις εκθέσεις. Δηλαδή, είναι καλό το να υπάρχουν ειδικέ προδιαγραφέ σε εθνικό επίπεδο, αλλά για μένα εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. αυτό θεωρώ ότι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων. Κατά τα άλλα, όσον αφορά στην καταγραφή των επιβατών ενός πλοίου, είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και από την άλλη να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Και άλλα δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Είναι σωστό ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μέσω του διαδικτύου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε πολλά στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις. Νομίζω πολύ σωστά το προτείνει αυτό η συγγήτρια. Και όσον αφορά το 1.11, πράγματι και εγώ ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, χρονική διάρκεια, πέντε ετών ή ακόμη και λιγότερο, όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Και τέλος, όσον αφορά αυτά που είπε κυρία Γιούτο, νομίζω είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα σκάφη μέχρι 24 μέτρα. Δηλαδή, κανόνες που θα έχουν και σχέση με την ασφάλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Βαντέλεν έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου σε θέματα ασφάλειας. Ε, και στις προδιαγραφές ε, για τους επιβάτες ε, και έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς την Κομισιόν. Δηλαδή, όταν πρόκειται για τον ορισμό των παραδοσιακών σκαφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα νέο ορισμό για τα παραδοσιακά σκάφη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι με αυτό το νέο ορισμό αποκλείονται σκάφη που μέχρι και το 65 ήταν επιβατικά σκάφη. Τα ιστορικά σκάφη, τα οποία τώρα, τα παραδοσιακά, τα οποία μεταφέρουν τώρα επιβάτες, δεν κατασκευάστηκαν ως επιβατικά αλλά ήταν ε, παγοθράφστες, ε, ρημουλκά, είχαν κατασκευαστεί για τέτοιου είδους ε, σκοπούς. Πρόκειται για τον ορισμό του 2295 και αν τον ε, εξακολουθούμε να το χρησιμοποιούμε αυτόν τον ορισμό, δεν θα υπάρχει πια πρόβλημα. Τώρα, η Κομισιόν γιατί θεωρεί ότι πρέπει ε, να υπάρχει νέος κανονισμός και να μην ισχύει πια αυτός του 2259. Λοιπόν- θα ήθελα, λοιπόν, να καλέσω τους προσκεκλημένους να πάρουν το λόγο. Ε, σας καλωσορίζω καταρχήν κύριε Σίμανς που είστε εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ στη σημερινή συνεδρίαση και σας δίνω το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας δίνετε την σύντομη αυτή δυνατότητα να εξετάσουμε αυτές τις τρεις ε, προτάσεις και να σας πω πως στις 19 Οκτωβρίου ε, ψηφίσαμε για το θέμα αυτό. Έχουμε και μια γνωμοδότηση ε, σχετική την οποία ε, σας έχουμε στείλει και θα χρησιμοποιήσω το χρόνο που έχω σήμερα εδώ για να μιλήσω περισσότερο για την έκθεση, για τις επιθεωρήσεις, την έκθεση ειρική γιατί είναι το θέμα το οποίο κατέχω καλύτερα. Να σας πω καταρχήν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό μέσω της προσπάθειας που γίνεται και μέσω του refit να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα είναι προσέγγιση ε, κράτους μέλους, εθνική δηλαδή, χωρίς όμως παρόλα αυτά να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα επιθεώρησης οποιοδήποτε αξιόπλου πλοίου και νομίζω πως σχετικά με το θέμα αυτό η οδηγία και αυτό είναι το σχόλιο μου ε, θα πρέπει να τονίζει ακόμα πιο πολύ τα τεχνικά σημεία τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια βελτίωση στο χώρο αυτό. Μία από τις προτάσεις για παράδειγμα η οποία γίνεται και στην οποία θα ήθελα να κάνω κάποια παραπάνω σχόλια. είναι η ομάδα επιρρογνωμόνων και για τα δικαιώματα των επιβατών αλλά και για την επιθεώρηση από το κράτος λιμένα. Καλό είναι αυτές οι δύο ε, επιτροπές να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε και ε, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές να έχουμε μια καλύτερη παρακολούθηση ε, αλλά και ε, εφαρμογή όλων όσων θα αποφασιστούν. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει προκύψει από τη συζήτηση είναι το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τους, τα επικίνδυνα σημεία όταν γίνονται, αυτοί οι, όταν γίνονται αυτές οι επιθεωρήσεις από το κράτος λιμένα. Νομίζω πως εδώ η, υπάρχει ένα αδύναμο σημείο, οπότε πρέπει να εστιάσουμε στο άρθρο 5, πρώτη παράγραφο, που λέει πως τα κράτη-μέλη πρέπει να συντονίζουν τις επιθεωρήσεις αυτές, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πως οι επιθεωρήσεις γίνονται αποτελεσματικά και αποδοτικά. Επίσης, έχουμε τον ορισμό των ρυθμιζόμενων ε, υπηρεσιών και επειδή πρόκειται εδώ για οδηγία, είναι πολύ πιθανό να έχουμε διαφορετικές ερμηνείες σε κάποια σημεία. Οπότε νομίζω πως καλύτερα θα έπρεπε να έχουμε έναν ανοιχτό ή έναν αναμειγμένο, ένα blended κατάλογο ε, αυτά ήταν τα σχόλιά μου και ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο που μου δώσατε, αλλά είχα αρκετά σχόλια όπως ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις. Προστασία δεδομένων, καταξουσιοδότηση πράκτης, ε, ενιαία θηρίδα. Οπότε ακόμα και τα σημεία για τους κοινωνικούς εταίρους που θέσατε κυρία Γιούτο. Οι προθεσμίες μεταξύ ε, και συχνότητα των επιθεωρήσεων. Ε, θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις και γι' αυτό σας δίνουμε το λόγο, κυρία Κουσίνσκα. Προέρχεστε από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Κοσένσκα. Συγγνώμη, Κοσένσκα. Good afternoon. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Ξέρω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο. Θα είμαι συντομότατη. Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν και όλη την Επιτροπή που εξετάζει από κοινού τις τρεις ε, εκθέσεις. Δεν είναι πολύ εύκολη η προσέγγιση. Όμως εφόσον ασχολούμεθα με την ασφάλεια των πλοίων, μπορούμε έτσι να διερευνήσουμε καλύτερα τις συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ διαφόρων νομοθετημάτων. Θα προσπαθήσω να διατρέξω τις ερωτήσεις. Αν λησμονήσω κάτι και τελειώσει ο χρόνος, να επαναλάβω εκ νέου ότι με τα χαράς να συζητήσω με τους ηγητές και τους σκιώδης ηγητές το θέμα πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες επί των τριών εκθέσεων. Ξεκινώ λοιπόν από την έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου. Πολλές τροπολογίες που πρότεινε η συγγήτρια είναι πολύτιμες. Κάποιες από αυτές πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Όπως ε, καθυστέρηση τη των στοιχείων πιβατών, αν θα πρέπει από 30 λεπτά να πάει στα 10 λεπτά. Το εξετάσαμε προσεκτικότατα, ετοιμάζοντας την πρότασή μας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είτε μιλάμε για 10 λεπτό είτε ημίωρο. Αλλά σε κάποια σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής παρατήρησα ότι το συντομότερο χρονικό διάστημα είναι προτιμητέων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν επιβληθεί αυτό θα επικρατεί σαφήνεια και προβλεψιμότητα για τους εμπλεκόμενους φορείς. Τι σημαίνει ένα δεκάλεπτο. Από ποια στιγμή μετράμε το δεκάλεπτο. Τώρα κολλάω σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά όταν μιλάμε για πολύ σύντομες χρονικές περιόδους είναι σημαντικό να επικρατεί απόλυτη σαφήνεια για όλους τους εμπλεκόμενους. Σημαντικότατο θέμα τώρα. Τα συστήματα πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθούν στην ενιαία θηρίδα. Παραδεχόμαστε ότι το σημαντικότερο και στόχος μας είναι να είναι εύρυθμο το σύστημα. Να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία. Εν την περίπτωση υπάρχει ο πειρασμός να παραπέμψουμε σε υπάρχοντα συστήματα. Να υπενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη επεξεργάζονται επί πάνω από εξαετία την χρήση εθνικών ενιαίων θηρίδων. Βλέποντας λοιπόν αυτό το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η οδηγία για την εφαρμογή αυτού, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί πλαίσιο το οποίο να είναι ούτως υπήν αιώνιο, να μην επηρεάζεται χρονικά. Εάν έχουμε απομονωμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένη διαδρομή, ο μακροπρόθεσμος στόχος να έχουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση με αναλόγια, ευρωπαϊκό σύστημα που θα επιτρέπει ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί η τροπολογία που αφορά τους επιβάτες που χρειάζονται ειδική βοήθεια, το δεχόμαστε αυτό, όσον αφορά αν θα είναι δύο χρόνια ή επτά χρόνια υποβολή των διαφόρων ε, εκθέσεων και αναφορών, αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε. Να πω ότι όσον αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη, βάσει πληροφοριών που απαιτούν περαιτέρω εξακριβώσεις και ελέγχους, και επαλήθευση συμμόρφωση. εκεί χρειάζεται κάποιος χρόνος. Και γι' αυτό αναφέρουμε έξι μήνες και όχι τρει μήνες. Ακούστηκαν διάφορα σχόλια που αφορούσαν το χρονικό διάστημα την υποβολή στοιχείων επιβατών. Η ε, κυρία Μοντέρο έθεσε ένα πολύ σωστό θέμα. το όριο των διαδρομών, γιατί 20 ναυτικά μίλια και όχι τις αποστάσεις του Σόλας. Αν συμπεριλάβουμε 20 ναυτικά μίλια, τότε 90% των δρομολογίων εσωτερικού που είναι σημαντικά θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Το προτείναμε αυτό για να έχουμε πληρέστερο πλαίσιο, να έχουμε μεγαλύτερη κάλυψη να καλύπτουμε διαδρομές που είναι σημαντικές για την ασφάλεια των επιβατών. Να καλύπτονται την οδηγία. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Τέιλορ για την εφαρμογή της νομοθεσίας, ελπίζουμε εμείς ότι αν διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογής, αν υπάρχουν λιγότερες παρανοήσεις για το τι πρέπει να γίνει από ποιον, αυτό διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας, που είναι και ο βασικός στόχος της προσέγγισης για το ΡΙΦΕΤ. Υπήρχε κάτι άλλο. Για τη συγκεκριμένη έκθεση. Αναφέρθηκε κοινωνική διάσταση. Ετέθη σχετικό ερώτημα. Δεν έχω κάποιο σχόλιο. Προσβλέπουμε στην παραλαβή των σχετικών τροπολογιών και μετά θα επιστρέψουμε. Υπόθηκε κάτι για την αναγκαία κατάρτιση των πληρωμάτων και τι, πώς αντιμετωπίζονται κατεπήγοντα περιστατικά και καταστάσεις ανάγκης. Το πλαίσιο της κατάρτισης υφίσταται. Αποτελεί κομμάτι του ελέγχου που κάνουμε για την καταλληλότητα του πλαισίου για τον επόμενο χρόνο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Για διασυνορική συνεργασία, πράγματι για εσωτερική ναυσιπλοεία για ατυχήματα που ίσως συμβούν σε διασυνοριακό πεδίο, ίσως δημιουργούνται προβλήματα. Στις θαλάσσιες μεταφορές η συνεργασία μεταξύ των ομάδων έρευνας και διάσωσης είναι εξαιρετική. Δεν είχαμε πολλές περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα. Ίσως να ήταν πιο περίπλοκη η κατάσταση έρευνας και διάσωσης, κυρίως σε επιχειρήσεις ξηράς, Εκεί χρειάζεται καλύτερη διαβίβαση πληροφοριών στους επιβάτες για να διευκολυνθεί η κατάσταση, αν προκύψει κάποια ανάγκη. Όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Αγιούτο, το ζήτημα της ασφαλείας των σκαφών και τα σχετικά πρότυπα, ένα σχόλιο για τις προδιαγραφές. Θέλαμε να παραπέμψουμε σε διεθνείς προδιαγραφές. Στην έκθεση για το Refit βάλαμε στοιχεία και στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν ακριβώς τη συμπεριφορά του ΣΥΠΗΝ, του χάλιβα και του αλουμινίου και των σχετικών σκαφών. Δεν θέλαμε όμως την πρόταση να αναφέρουμε προδιαγραφές που δεν υπάρχουν ακόμα σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό κάποια είδη σκαφών δεν καλύπτονται ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή θα υπάρξουν συμπεφωνημένε διεθνεί προδιαγραφέ δεν θα είναι εφικτό να καλυφθούν από την οδηγία. Άλλο ερώτημα αφορούσε τα λευτικά σκάφη. Υπάρχει μια διεθνή σύμβαση που ισχύει για τα λευτικά σκάφη. Δεν λειτουργεί απολύτως καλά. Εφόσον προσπαθούμε να διατυπώσουμε την ομοθεσία το να εντάξουμε πλήρως τα ληφτικά σκάφη στο πεδίο εφαρμογή οδηγία θα ήταν κάτι ανέφικτο. Διότι θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε σε σημαντικό βαθμό το πεδίο εφαρμογή του νομοθετήματο. Του του λεχθέντο. Σα διαβεβαιώνω ότι συνεργαζόμαστε στενά με του συναδέλφου τη DG Mare και θα διαβιβάσουμε τα ερωτήματά σα σε αυτού. Α, ναι, ναι. Υπήρχε και το άλλο για τα παραδοσιακά σκάφη και τις προδιαγραφές. Πώς ορίζονται τα παραδοσιακά σκάφη. αναφερόμαστε σε επιβατηγά σκάφη που ναυπηγήθηκαν πριν το 1965 και όχι σε σκάφη που αργότερα μετετράπησαν σε επιβατηγά σκάφη. Θέλαμε να έχουμε ένα νομοθέτημα που έχει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη. Δεν θα ήταν επωφελές για κάποιον να περιοριστεί αυτό το πεδίο, διότι συζητούμε την ασφάλεια των σκαφών. Ίσως ε, να θεωρείται από κάποιους ότι μερικώς, πώς να το πω, περιορίζουμε τον ορισμό των ιστορικών σκαφών και έτσι το πεδίο εφαρμογή ε, διευρύνεται. Τώρα θα δούμε Επίσης, ε, στην έκθεση της κυρίας Αγιούτο γίνεται λόγος για επιπρόσθετες εξηγήσει ε, σχετικά με τις ε, προδιαγραφές. Λοιπόν, ε, οι διεθνώς συμφωνημένες προδιαγραφές. Ε, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να αποδώσουμε σημασία σε ορισμένα άλλα θέματα, όπως τα ιστιοπλώα, τα ιστιοφόρα ε, και τα τέντερ, τα μικρά σκάφη. Μισό λεπτό να δω αν ξέχασα κάτι, κάποια σημαντική ερώτηση σχετικά με τις προδιαγραφές. Νομίζω αυτά τα είπα. Το θέμα των ε, σκαφών ε, από αλουμίνιο τέτοια επανειλημμένα. Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους γιατί ε, κατατίθεται αυτή η πρόταση είναι ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι τα σκάφη από αλουμίνιο που υπάρχουν αυτά θα καλύπτονται από την οδηγία και στόχος μας είναι να είναι εξίσου ασφαλή όπως και αυτά από χάλιβα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία που αφορούν ε, στην αυπήγηση σκαφών ε, από αλουμίνια. Μας ενδιαφέρει η ασφάλειά τους να είναι ίδια όπως και στα άλλα. Ο κύριος Ρουκέ πολύ σωστά είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ λεπτό θέμα στο θεματολόγιο του Συμβουλίου αλλά επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο τρισμερής διάλογος, ίσως ε, να μην πρέπει να τα σχολιάσω αυτά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω και έτσι κι αλλιώς ε, έχω προκαιρού σπαταλήσει το χρόνο που είχατε προβλέψει για μένα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Ήταν σημαντικό να δοθούν απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις που ετέθησαν τους βουλευτές της Επιτροπής μας. Εντάχει, να δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον καθένα από τους ηγητές μας, διότι πιστεύω ότι και αυτοί επίσης ε, θα έχουν ίσως κάποια ερωτηματικά. Σύμφωνα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν γέννη πιστεύω ότι συμφωνούμε. Πράγματι υπάρχει μια συμφωνία και συμφωνούμε όλοι ότι όσον αφορά της κατεξοδότηση πράξης ε, πρέπει να είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα. Εξάλλου είναι απαραίτητο να υπάρχει προστασία δεδομένων ε, και αυτό που παίζει επίσης ρόλο είναι ότι ετέθησαν ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με τα δεδομένα ε, εμείς συμφωνούμε ότι όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται σε ένα μητρό και σε περίπτωση ατυχήματος να γνωρίζουμε πολύ καλά ε, κατά πόσον ε, υπήρχαν επιβάτες και ποιοι ήταν ακριβώς ε, οι επιβάτες στα σκάπη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε ταυτοποίηση των ατόμων σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης με, την, με το Ευρωπαϊκό Μητρό Πρέπει να σας πω πως εδώ θα πρέπει να υπάρχει δια... συνδεσιμότητα με τα εθνικά μήτρωα. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε πως εδώ και έξι χρόνια έχουμε τα εθνικά και άρα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκό. Μα δεν λειτουργούν. Είχαν έξι χρόνια στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη για να τα θέσουν σε εφαρμογή, για να συντονίζονται τουλάχιστον μεταξύ τους έτσι ώστε ο κλάδος να έχει την εντύπωση ότι τα πράγματα πάνε καλά, αλλά για μια φορά ακόμα αυτά τα εθνικά μητρώα μετά από έξι χρόνια δεν λειτουργούν. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγα ήταν πως θα πρέπει να βελτιωθούν και είπα πως αποτελεί πρόκληση γιατί θα πρέπει πρώτα τα εθνικά μητρώα που δεν λειτουργούν να βελτιωθούν και μετά ενδεχομένως στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε και ένα ευρωπαϊκό μητρό, όχι ως σκέψη να το στην τρέχουσα οδηγία. Για τα 30 λεπτά και κατά πόσο αυτά θα γίνουν 10 λεπτά. Κοιτάξτε, τα όσα είπε η Κομισιόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να μειωθούν και μας είπε προσέξτε γιατί από τη στιγμή που μειωθούν δεν θα έχουμε προβλεψιμότητα. Μα από πότε ξεκινάει κανείς να μετράει είτε 30 λεπτά είτε 10, το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε από ποια στιγμή αρχίζει να τρέχει το ρολόι. Σας παρακαλώ πολύ, ε, συνάδελφε, πρέπει να τελειώνετε. Ναι, τελειώνω, αλλά πρέπει να σας πω πως θα πρέπει και εδώ τα πράγματα να είναι ξεκάθαρο. Για τα 10 λεπτά τα ίδια προβλήματα έχουμε είτε είναι 30, είτε είναι 25, είτε 10. Άρα λοιπόν Νομίζω πως απαντήσαμε στις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι για το πώς θα χειριστούμε και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιούτο. Ε, δεν έχω χρόνο, λοιπόν θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Φώστερ προφανώς ε, και θα πρέπει να ε, εναρμονιστούμε με τις προδιαγραφές του IMO ε, χωρίς να είμαστε πιο περιοριστικοί. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις γκρίζες ζώνες, επ' αυτού συμφωνούμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα του αλουμινίου. Είναι αλήθεια ότι στην οδηγία δεν ορίζεται το θέμα του ισοδύναμου. στο παράρτημα 1, κεφάλαιο 2, εκεί αναφέρονται οι προδιαγραφές για το ποια τμήματα μπορούν να είναι από αλουμίνιο. Ε, Άρα δηλαδή το να αποκλείσουμε το όλο θέμα του αλουμινίου είναι ε, σαν να θέλουμε να παρακάμψουμε το θέμα του ισοδύναμου. Ε, κατανοούμε όλο αυτό το θέμα που έχει σχέση με τη Γαλλία, ότι είναι απαραίτητο να προστατευτεί ένας βιομηχανικός κλάδος, θέσει εργασία. Δεν θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτό. Γι' αυτό ας βρούμε από κοινού μια λύση, γιατί πράγματι στόχος είναι να υπάρχει ασφάλεια και νομίζω ότι αυτό το θέλουμε όλοι και όλοι πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση ο κ. Ρικέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές. Άκουσα μεγάλη προσοχή. Για να μην χρονοτριβώ, να πω δύο πράγματα. Για την κυρία Μοντέρα, ο, ο χαρακτήρας, ο μη εποχιακός δεν οδηγεί σε παρεκκλήσεις η φόρτωση, η υπερφόρτωση κατά σεζόν κλπ. δεν του οδηγεί σε απαλλαγή. Έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση των δύο μηνών για να μην του εμποδίζουμε στις εργασίες του. Είναι πιο εύκολο να, μην, να γίνονται έλεγχοι όταν δουλεύουν 360 μέρε το χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ειδική, ειδικός έλεγχος όταν υπάρχει ασύμμετο χαρακτήρα στην κυκλοφορία. Κύριε Τέλερ, όσον αφορά το προσωπικό, στις επιθεωρήσεις εξετάζονται όλα τα θέματα προσωπικού και θα πρέπει να συμπληρώνεται ε, στο ημερολόγιο το θέμα ότι το προσωπικό πρέπει να κάνει εξηγήσει και πρέπει να υπογράφονται αυτέ οι είσοδοι στο ημερολόγιο πλοίου. Η κατάρτιση δεν είναι θέμα τη επιθεώρηση, επαληθεύει όμω η επιθεώρηση ότι γίνονται ασκήσει και η κατάρτιση. Από αυτή την πλευρά λοιπόν ε, δεν χρειάζεται συμπληρωματική ε, διατύπωση λαμβάνω υπόψη τα υποθέντα, κυρίως αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Οικονομικό Κοινωνικό. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, γίνονται οι τροπολογίες κατά ε, έκθεση. Προθεσμία είναι 9 Μαρτίου για την υποβολή τροπολογίων για τις εκθέσεις. Μεσημέρι. Συνεχίζουμε, αφού ευχαριστήσω τους συζητητές μου, με τους χρηματοστατικού κανόνε που εφαρμόζονται για τον γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή στο σχέδιο προ εξέτηση στην Επιτροπή Προπολογισμών και τη Συνταγματική Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ο κ. Βιμ Βαντεκάμπ είναι ο εισηγητή ε, για να παρουσιάσει την σχετική γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως ε, θα πρέπει λιγάκι να δούμε τον ε, προγραμματισμό της ε, συνεδρίασης γιατί τρεις εκθέσεις σε μία ώρα δεν φτάνει και εγώ είχα και την εντύπωση ότι θα ήθελα να τοποθετηθούν και οι σκιώδεις ηγητές. Μπας περιπτώσει, πάμε τώρα στον κανονισμό Omnibus, έτσι λέγεται ο κανονισμός αυτός, πρόκειται για τους, ε, για τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτό ε, θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. Η Επιτροπή Μεταφορών δρομολόγησε τη διαδικασία με βάση το άρθρο 55 για την αλλαγή τροποποίηση του σχετικού κανονισμού. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για αυτό το θέμα και είμαστε αρμόδιοι να γνωμοδοτήσουμε. Οι επιτροπές Τραν, η Ρέγγι, η Επιτροπή Επασχόλησης, η Επιτροπή Περιφερειών ε, και αυτές οι επιτροπές έχουν κάποιες αρμοδιότητες. Κυρία Πρόεδρε, στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου ασχολούμαι κυρίως με την ε, με το εργαλείο της μικτής χρηματοδότησης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μείγμα κυρίως αναφορά αφορά τις ε, δαπάνες για τα έργα υποδομής. Μας ενδιαφέρει να τροποποιήσουμε το σχετικό κανονισμό. Επίσης, τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και σε άλλα τμήματα. Αυτό όμω δεν το περιλαμβάνω στη γνωμοδότησή μου. Αν οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν και άλλες ε, τροποποιήσεις, θα έλεγα να τις κάνουν μέσα από την Επιτροπή Κόντ ή από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ή από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Εγώ έχω προετοιμάσει μία σειρά τροπολογιών, νομίζω το είδατε αυτό. Ε, η πρώτη ομάδα τροπολογιών είναι υπαριθμών 1 έως 4 και εκεί πρόκειται για την εξήγηση κάποιων τεχνικών θεμάτων στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά δεύτερον, ε, θέλουμε να επιβάλλουμε στην Επιτροπή την υποχρέωση αναφοράς, ε, κυρίως όσον αφορά κατά την εφαρμογή του μικτού χρηματοδοτικού εργαλείου. Γιατί νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί κατά τα επόμενα έτη. Η τρίτη ομάδα των τροπολογιών ε, πρόκειται για την επέκταση της ε, μικτής χρηματοδότησης και νομίζω ότι οφείλουμε ε, στον χρηματοδοτικό τομέα να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν ε, περισσότερα εργαλεία γίνεται. Ε, γνέριζουμε ότι υπάρχει αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών και γνωρίζουμε ότι οι συνεργασίες δεν λειτουργούν πάντα αποτελεσματικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Και αν τελικά ε, στο εργαλείο της μικτής χρηματοδότησης ε, ε, παραμείνει κάτι και δεν χρησιμοποιηθεί, αυτό θα πρέπει να επανέλθει στο ΣΕΦ, στις επιδοτήσεις και δεν θα πρέπει να χαθεί κάπου στο γενικό προϋπολογισμό, στο ΕΦΣΙ, στο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την έκθεση που είναι πραγματικά άριστη και αυτό με παραξενεύει βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω πως Πρέπει να δούμε καταρχήν ε, τι γίνεται με το μηχανισμό ε, Connecting Europe. Για το τμήμα Α του προπολογισμού θα απευθυνθούμε κατευθείαν στην Επιτροπή Προπολογισμού και νομίζω ότι ο νέος κανονισμός αυτό δεν το επιτρέπει πια. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να καταθέτουμε ως μέλη μιας επιτροπής τροπολογίες προσωπικές σε άλλη επιτροπή. Αυτό δεν λέει ο καινούριο κανονισμός. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία σε ποιο τμήμα βρισκόμαστε. Το τμήμα 1α και α του τακτικού προπολογισμού είναι αυτό που απασχολεί, μάλλον που αναφέρεται στις μεταφορές. Άρα λοιπόν εμείς πια προσωπικά δεν έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε τροπολογίες στην Επιτροπή Προπολογισμού. Αφενός αυτά. Αφετέρου. Συμφωνώ πως το blending είναι ένα θέμα το οποίο είναι ύψης της σημασίας και το γεγονός πως μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία πραγματικά τα ενισχύει σε μεγάλο βαθμό. Το ζήτημα είναι να απαντήσουμε στην εξής ερώτηση. Πού θα βρούμε τα κονδύλια για να ενισχύσουμε ε, το πακέτο Juncker. Είτε στο Connecting Europe, το οποίο είναι ένα ταμείο και τα ταμεία δεν ανήκουν στο γενικό προϋπολογισμό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω πως στο γενικό προπολογισμό έχουμε κάποια ταμεία που είναι τα περιφερειακά ταμεία, τα οποία είναι ταμεία ανταγωνιστικότητας και ταμεία για τα κράτη συνοχής. Αυτά τα λέω για να σας τα και να με παρακολουθείτε. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μπουν ε, στο μηχανισμό blending και να στηρίξουν με τον τρόπο αυτό και το εύση. Όμως ο κανονισμός που διέπει αυτά τα ταμεία ε, και κυρίως το ΕΤΠΑ δεν το επιτρέπει. Και αν δούμε τι γίνεται με το Ταμείο Ανταγωνιστικότητα, γιατί ίσω εκεί θα έπρεπε περισσότερο να εστιάσουμε, είναι πω δεν μπορούμε να αλλάξουμε του κανόνε που επηρεάζουν ε, τις μεταφορές και κυρίως το σύνδεσμο που δίνουμε εμείς με την ανταγωνιστικότητα. Άρα λοιπόν λόγω οικονομικού κανονισμού εδώ για τα ταμεία αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή blending. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποια κονδύλια εκτό τακτικού προπολογισμού, κάτι το οποίο περιπλέκει την κατάσταση. Το δεύτερο, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι πρέπει να απαιτήσουμε εμείς και δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως κανόνα ή ως κάποιο εκτιμώντας να απαιτήσουμε ότι όταν συζητάμε ε, από όσους υποφάλουν υποψηφιότητες για το επενδυτικό ταμείο Juncker είτε για κάποιο άλλο ταμείο ε, να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση που η ΕΤΕ δεν αναλαμβάνει το κίνδυνο πρώτης απώλειας. Οπότε, θα μου πούνε σε τι εξυπηρετεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός που είναι ε, είναι ε, ευρωπαϊκά χρήματα του φορολογούμενου ε, να ε, βάζει στη διάθεσή μας τέτοιου είδους κονδύλια μέσω του πακέτου Juncker έτσι ώστε να έχουμε εγγύηση πρώτης απώλειας και μετά να μην το δέχεται η ΕΤΕ με αποτέλεσμα να πρέπει να το μοιραστούμε με άλλους επενδυτές. Οπότε, πώς μειώνουμε τον κίνδυνο ε, μέσω επιδοτήσεων. Αν όμως αυτή τη στιγμή λέμε πως μειωνουμε τον κινδυνο μεσω επιδοτησεων αν ομως αυτη τη στιγμη λεμε πως προκειται για επιδότηση πλάτες δηλαδή ε, μόχλευση, ερεσιμότητα, Οκ, okay, αλλά θα πρέπει και η ΕΤΕ αυτή την, ε, το κίνδυνο πρώτης απώλειας να τον αναλαμβάνει έτσι ώστε να χρηματοδοτεί επιπλέον ε, πράξεις. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κράμερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Έλαβε υπόψη πολλά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης υποχρεώσεως ενημέρωσης. Έχουμε το Ταμείο Γιούνκερ. Υπάρχουν δισεκατομμύρια, αλλά δεν υπάρχει κάποια ανάλυση αυτού. Όμως ελήφθη απόφαση να επεκταθεί το Ταμείο. Δεν είναι μόνο θέμα των χρημάτων, αλλά πού πηγαίνουν τα χρήματα Πώ αποδεικνύεται η επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται με την προστασία του κλίματο με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, Χρειάζεται μια ανάλυση για να βλέπουμε κατά πόσο πετυχαίνουμε του στόχου. Υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα, υπάρχουν όμω και πολλά αρνητικά παραδείγματα και γνωρίζουμε καμιά φορά ότι τα χρήματα επίση μπαίνουν σε κάποιε σκοτεινέ διαβλούς. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με τα χρήματα για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και την ιδέα του κυρίου Βαντεκάμπ για μεικτή χρηματοδότηση, θα να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ακούγονται πολλά. Υπήρξε κάποια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Άκουσα ή κάτι τέτοιο που γίνεται στην Ελβετία. Και η Ελβετία μου είπαν όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Όταν ρώτησα του Ελβετού για τη σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Όταν πηγαίνει καλά ένα έργο, ε, χρηματοδοτεί ο δημόσιο τομέα Λοιπόν, αυτή η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη Γερμανία κατά 90% ήταν πιο δαπανηρέ. Όταν, όταν συμμετείχε μόνο το κράτο, αυτά τα έργα ήταν 90% πιο ακριβά από ότι όταν υπήρχε σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία για να ξέρουμε αν κινούμεθα προ σωστή κατεύθυνση. Ξέρω πολλά για τη διαφθορά. Στην Ισπανία πριν από 10 χρόνια ασχολήθηκα με αυτό. Λοιπόν, βλέπαμε τελικά ότι υπήρχαν πολλά, πολλά φορτηγά που κυκλοφορούν στις εθνικές οδούς. Φαρά τις προσπάθειες για το αντίθετο. Λοιπόν, και υπήρχε πρόβλημα με το θέμα της ιδιωτικοποίησης των αυτοκινητοδρόμων κυβερνήσεως Ασνάρ, τότε στην Ισπανία. Εκείνοι που έκαναν την ιδιωτικοποίηση ε, χρεοκόπησαν αυτοί που συμμετείχαν. Και το κράτος έπρεπε να επαναγοράσει για 5 δισεκατομμύρια ευρώ τους αυτοκινητοδρόμους. Γιατί ε, και πώς, μέσω συμβάσεως. Τα κέρδη θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Δεσμεύτηκε όμως το κράτος να καλύψει τα ελλείμματα και αγόρασε για 5,5 το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ισπανία, το Ισπανικό κράτο. Ο όμιλο που ιδιωτικοποίησε το αυτοκινητοδρόμους αποτετείται από εταιρείε, από επιχειρηματίες ε, των ε, οικοδομών που θεωρούσαν ότι θα ήταν επικερδές να ιδιωτικοποιηθούν οι αυτοκινητόδρομοι. Όμως δεν αρκούσαν τελικά τα διόδια για τη χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων τον Όμιλο δεν τον ενδιαφέρει η χρηματοδότηση μέσω των δίων, μόνο η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Και τελικά χρεοκόπησε τότε στην Ισπανία ανά χιλιόμετρο κοστίζε το διπλάσιο από ότι στη Γερμανία αυτοκινητόδρομος. Αυτό ήταν παράλογο, έτσι δεν είναι. Στην πραγματικότητα όμως ήταν καλυμμένη διαφθορά που έλαβανε χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να, να βλέπουμε από κοντά Ε, όταν ο κύριος Μπερλουσκόν ήταν στην κυβέρνηση, υποτίθεται είχε υποσχεθεί στην μαφία να κάνει κάποιο αυτοκινητόδρομο στη Μεσίνη. Και μετά όμως διαγράφει αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ε, στην Οντουρίν ε, έχουμε δύο ε, TGV παραπάνω που θα ε, υπάρχει αυτή η σύνδεση. 26 δις θα στοιχήσει αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλα αυτά να γίνουν και η Κομισιόν οφείλει να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο το οικονομικό και να λέμε όλα πάνε τέλεια. Ε, δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι η έκθεση του ΔΥΜ είναι πάρα πολύ καλή και οφείλουμε να παρακαλέσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε τι πληροφορίε. Τελικά τι έγινε με αυτό το πρόγραμμα του κ. Γιούνκερ στον τομέα των μεταφορών. Ποια προγράμματα συμπεριληφθήκαν, ποια απορρίφθηκαν. Για τίποτα δεν έχουμε καμία αιτιολογία και νομίζω ότι ω κοινοβούλιο αυτό είναι άδικο. Οφείλουμε τουλάχιστον να ενημερωνόμαστε. Βλέπω ότι ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν νέφει καταφατικά. Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Και αν αυτό το, ε, η κίνηση του να ανέβει καταφατικά μεταφραστεί και σε πράξεις, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ και Κράμερ. Η κυρία Κιλώνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Βαντερκάμπ. Τον ευχαριστούμε για τη γνωμοδότησή του. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού για τη χρηματοδότηση. Έχω και εγώ παρόμοιες ανησυχίες. Κατά πόσο οι μηχανισμοί χρηματοδότησης εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πάντα ανησυχούμε για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όποτε το κουβεντιάζουμε. Τελικά όμως στην πράξη δεν κάνουμε πολλά για να αυξήσουμε τις δυνατότητες επιβίωσής τους. Όταν μιλούμε για εργαλεία όπως το Ταμείο Στατικικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι σπάνιο μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το πρόβλημα, να το εξετάσουμε σοβαρά. για να μην επικρατούν άδικε συνθήκε στην αγορά. Δεύτερον, ε, ποιε είναι οι συνέπειε χρηματοδότηση. Αν έχετε επισκεφθεί κάποια εκδήλωση εκτός κοινοβουλίου πρόσφατα με θέμα της μεταφορές, θα παρατηρήσατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, για την ιδιωτικοποίηση κλπ. Το ερώτημα όμως είναι τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρηματοδοτεί παλιωμοδίτικα προγράμματα όταν η τεχνολογία αλλάζει ριζικά. Και όταν υπάρχει ταχεία ανανέωση στον τομέα. Εγώ φοβάμαι ότι δεν δίνουμε με σωστό τρόπο τα σωστά έργα ε, τη χρηματοδότηση. αρκετές φορές δίνονται πόροι για τη μείωση των εκπομπών της κυκλοφορίας. Συνάδελφοι, εγώ θα εξακολουθώ να πολεμώ για τη σωστή χρήση των πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίλσεν είναι ο επόμενος ομιλητής. Tack κοιτάξτε, εγώ είμαι στην Επιτροπή ΡΕΓΙ. Τα κονδύλια από το Περιφερειακό Ταμείο υποτίθεται θα ε, εμβαστούν, θα μεταφερθούν στο ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Για να γίνει αυτό πρέπει να οριστούν οι κανόνες. Και υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που ισχύουν για το Περιφερειακό Ταμείο. Δηλαδή, σε περίπτωση υποδομών στρατηγικής σημασίας γίνονται επενδύσεις και οι περιφέρειες έχουν προτεραιότητα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Επίσης, ε, οι αρχές ε, θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικά. Δεν μπορούν να γίνουν όλα τόσο απλά. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ε, τα οποία θα συζητήσουμε στην Επιτροπή Περιφερειών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσω να μας απαντήσει. Κύριε Μαρίν, πείτε μας. Καταρχήν καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και να σας πω για τις ερωτήσεις που έγιναν, για τα όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Μπορείτε να απαντήσετε και μετά ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Και να σας πω ότι όντως Έχετε κάνει αρκετές ερωτήσεις και πρέπει να σας πω πως η τροπολογία η οποία προτείνεται οι τροπολογίες μάλλον είναι αρκετά καλές για μας και θα τις λάβουμε δεόντως υπόψη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συμβολή σας στη συζήτηση. Uh, uh, Όσο δε για το θέμα του blending, νομίζω ότι η προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα εδώ ε, περιορίζεται στο Connecting Europe ε, Facility. Και νομίζω ότι η συζήτηση για blending με τα ταμεία συνοχής και τα διαφορετικά ταμεία είναι ένα επόμενο κεφάλαιο της συζήτησης. Ίσως εκεί που έχουμε τις κοινέ διατάξεις και το σχετικό κανονισμό. Κάτι το οποίο βεβαίως συζητήθηκε στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου, του Omnibus με την DigiRegio, η οποία είναι και αρμόδια, αλλά καταγράφω παρόλα αυτά που η συζήτηση ξεπερνά ε, τα, τον περιορισμό του blending μόνο με το Connecting Europe Facility. Επίσης, Επίσης, νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα εδώ για να απαντήσω και στα όσα είπατε για το σημείο κίνησης γιατί εδώ ε, έχουμε την ε, ΕΤΕ και την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ που για τον κίνδυνο πρώτης απώλειας είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει να κάνει κυρίως με την τιμολόγηση και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε ε, σε μια τέτοιου δομή να χρησιμοποιούμε το ΕΕΦΣΙ, ε, το Ευρωπαϊκό δηλαδή Επενδυτικό Ταμείο, ως μια πλατφόρμα που θα βοηθά τη στιγμή της πρώτης επένδυσης. Τώρα για την προσθετικότητα, ε, για την αιρεσιμότητα δηλαδή, ε, νομίζω ότι το σχετικό θα συμπεριληφθεί στην πρόταση για το FC2. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο νομοθετικό πλαίσιο του ε, FC που προετοιμάστηκε πριν από 1,5 χρόνο, αλλά ως παράλληλη συζήτηση με τη συζήτηση που τρέχει για την κανονισμό Omnibus είναι τα όσα θα συμπεριλάβουμε στο FC2, όπου εκεί η αιρεσιμότητα έχει ήδη συμπεριληφθεί στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα κλείσω λέγοντας πως το θέμα των καλύτερων και πιο διάφανων ε, υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και αναφοράς η πρόταση που έκανε για το FC2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα ζητήματα που έχετε θέσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Επενδυτική Επιτροπή να λαμβάνει μια μεμονωμένη απόφαση για κάθε υποψηφιότητα ή πρόταση που υποβάλλεται μέσω του ΕΦΣΥ και βεβαίως η αναφορά να γίνεται και στο κοινό με πιο διάφανο τρόπο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρίν. Ο εισηγητής μας ε, μπορεί να σχολιάσει. Ik ε, wil hartelijk danken voor de zeer... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις συζητητές οι οποίοι πραγματικά παρακολούθησαν αυτή τη γνωμοδότηση δική μου ε, με επικοδομητικό τρόπο. Άσκησαν βέβαια κριτική. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ε, ζήτησε συγγνώμη, δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αν είχε έρθει εδώ θα είχε ασκήσει και εκείνη κριτική. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, για να απαντήσω πρέπει να μελετήσω. Θα τα μελετήσω και αυτή είναι η δουλειά μου που πρέπει να κάνω και θα επανέλθω. Ε, και για αυτά προς ο κ. Ρουκέ και ο κύριος ε, Νίλσον. Ε, βασικά μου έδωσαν έτσι τροφή για σκέψη και περισυλλογή. Και η Κομισιόν είπε ότι υπάρχουν θέματα που δεν αφορούν τη Γενική Διεύθυνση μου, αλλά ίσω τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγι ή αν θέλετε γενικά το Ταμείο συνοχή. Συνάδελφε Ρικέ, Μάρκους Πίπερ ε, και κύριος ε, Νίλσεν, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ένας από εκείνους οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα να τα βάλουν μαζί. Είμαι αρκετά γενναιόδωρο σε αυτό. Ας πούμε, παράδειγμα, πήγαμε στη Ρουμανία και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώ εκεί δεν ε, ε, γίνεται σωστή απορρόφηση των κονδυλίων για τις μεταφορές. Κάπου έχουν κολλήσει τα κονδύλια. Και ο κύριος Νίλσον έχει δίκιο. Αυτό είναι ένα θέμα ουσίας. Δεν ξέρω αν μπορώ κάπως να το λύσω, αλλά ο κύριος Ρικέ λέει Ταμείο Συνοχής και Blending. Αυτό θα πρέπει να είναι κάπως ε, φυκτό. Και ο πρώτος ε, κίνδυνος ε, δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί υπάρχει το Ταμείο ΕΦΣΥ, υπάρχει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακριβώς για να αντασφαλίζονται αυτοί οι κίνδυνοι. Και ο επενδυτής είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Ακούω ε, πολλούς να διαμαρτύρονται ότι τελικά αυτή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει γίνει εμπορική τράπεζα. Αν όμως το βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Ε, κάτι δεν πάει καλά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ιερό τέρας εδώ στο Κοινοβούλιο. ότι αντιμετωπίζουμε όπως τον κύριο Γιούνκερ. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο κύριος Κράμερ τοποθετήθηκε στην υποχρέωση αναφοράς και εγώ το στηρίζω αυτό. Ε, το βρίσκω πραγματικά όμως δυσάρεστο το ότι τα ΣΔΙΤ αυτές οι συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προχωράνε τόσο αργά και το ότι ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα συνταξιοδοτικά ταμεία και αυτό το βρίσκω κρίμα. Όσον αφορά τη διαφθορά, θα επανέλθω από αυτού. Κάτι θα έχω να πω. Όσον αφορά τώρα στις ε, μικρομεσαίε επιχειρήσεις, το είπαν και οι συνάδελφοι ότι πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές φορές εύκολα λέγονται πράγματα, ότι εντάξει να κάνουμε κανόνες, δύσκολα γίνονται όμως. Ε, υπάρχουν ε, προγράμματα τόσο μεγάλα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν το ρόλο, κάποιο ρόλο στις υπεργολαβίες, αλλά όχι ως κομβικές επιχειρήσεις. Θα το ξαναδώ λιγάκι, αλλά δεν νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο blending ε, και η Κομισιόν θα το δει λιγάκι το θέμα και κάτι θα έχει να πει. Και αυτή όλη σχέση ε, με τις ε, υποδομές, αν θέλετε, η ψηφιοποίηση, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Η κυρία Κίλον έχει δίκιο. Μπορεί κανείς να συνδυάσει τις ε, σύγχρονες με τις ε, παλαιές υποδομές. Αλλά ξέρετε αγαπητέ συνάδελφοι, τελικά όμως μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά. Για να φτιάξουμε έναν δρόμο χρειαζόμαστε απλά άσφαλτο. Συνάδελφε Νίλσον, εγώ είμαι ένας από εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θέλω να συνδυάσω όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή Ρέγγι ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως τα κάνουν μόνες τους απομονωμένα. Ευχαριστώ κύριε Βήματα Καμ. Προθεσμοί για τροπολογίες είναι η 7η Μαρτίου το μεσημέρι στις 12. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με ένα τελευταίο σημείο, πολύ ενδιαφέρον. Κοινή συζήτηση ψηφιακή τεχνολογία στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και ευρωπαϊκέ προθεγραφέ για την εφαρμογή του κανονισμού. 1025-2012, σχέδιο γνωμοδότηση για τι επιτροπέ ΙΤΡΕ και ΙΜΚΟ. Θα αφήσω το λόγο στον εισηγητή μα, στον κύριο Τεβίνσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Σήμερα Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις μπροστά μας. Σχετίζονται με διαφορετική ανακοίνωση, όμως έχουμε έναν κοινό στόχο και κοινή προσέγγιση για την εφαρμογή της ψηφιακής ενίας αγοράς, όπως αποκαλείται. Ψηφιοποίηση είναι το ένα και το άλλο είναι τυποποίηση, το άλλο θέμα. Τα δύο αυτά θέματα θεωρώ ότι αποτελούν σημαντική συμβολή για τη δημιουργία μιας ολοκληρω... ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις που απαιτούνται και για καινοτομία και για υποδομές και θα βοηθήσει αυτό στην ανάπτυξη αντίστοιχων προτύπων. Και χρειάστηκε η αναγκαία κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, προετοιμασία του. για το μεταφορικό τομέα. Είναι στην πρώτη γραμμή ο τομέας των μεταφορών θα έλεγα. Όσον αφορά την καινοτομία στο ψηφιακό τομέα. Όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ήδη είχαμε μια έκθεση για την ψηφιακή αγορά ε, και τις μεταφορές. Η τρίτη γνωμοδότηση κυλών ήταν όπως θυμάμαι. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Το ζήτημα είναι πώς θα προσεγγίσουμε το ζήτημα, τι πρέπει να γίνει ούτω ώστε να συμβούν αυτά που πρέπει. Θα εξετάσω κάθε θέμα ξεχωριστά. Πάω στην τυποποίηση τώρα και τις προδιαγραφές. Να τονίσω δύο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ευφυείς μεταφορές ανήκουν στις υπηρεσίες που αναδύονται μέσω της τυποποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας σε πέντε βασικούς τομείς. Περιγράφει τους τομείς. Κυβερνοασφάλεια, νεφο, υπολογιστή στο διαδίκτυο των πραγμάτων, 5G και τα big data. Συμφωνώ, αλλά βλέπω δύο στοιχεία βασικά τα οποία δεν θα πρέπει να λησμονηθούν επί των οποίων πρέπει να στεφτούμε. Ευφύς δεν περιορίζεται στις μεταφορές αυτό, αλλά συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίε. όπως ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων και νέα κινητικότητα. Πρέπει αυτά να προωθηθούν και να αναπτυχθούν. Δεν αφορά μόνο τις μεταφορές αυτές καθ' και τις υποδομές, μιλούμε για κάτι που τίνουμε να λησμονούμε. Υπηρεσίες και τίνουμε να ακούμε τις απόψεις μεγαλύτερων φορέων της αγοράς και τουριστικών φορέων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Συνήθως αυτό αποτελεί δικαιολογίες και συνήθως τα εμπόδια αφορούν την υλοποίηση της νομοθεσίας. Δεύτερον, ανεξάρτητα από την ευφυΐα που διακατέχει τις μεταφορές, είναι θέμα υποδομών η μεταφορά τα συνδεόμενα αυτοκίνητα απαιτούν ανάπτυξη επικοινωνίας πέμπτης γενιάς 5G. Αλλά εξαρτώμεθα κατά πολύ και από τα εναλλακτικά καύσιμα, εναλλακτική ενέργεια τα νέα αυτοκίνητα. Άρα χρειάζεται να υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Αν δείτε ποια είναι η τωρινή κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οχήματα εναλλακτικά. Το θέμα είναι η μορφή των υποδομών, αν είμαστε έτοιμοι. Και η απάντηση κατά την άποψή μου είναι όχι, δεν είμαστε έτοιμοι χρήση νέων, νέου τύπου οχημάτων. Και είναι και θέμα διαλειτουργικότητας. Ε, βλέπω τι συνέπειες πρέπει να εξεταστούν. Πρέπει να προωθήσουμε ανοιχτές προδιαγραφές. Να μην εμποδίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τροπή, να προωθήσει τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Για να μην εφαρμόζουμε σε δεκαετία μη ευρωπαϊκές προδιαγραφέ. Πιο εύκολο να το πει κανεί, παρά να το κάνει βέβαια. Αλλά λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε πολύ ισχυρού ανταγωνιστέ. και το πώ μόνοι μα αποδυναμωνόμεθα, αυτό δεν θα το θεωρούσε ότι είναι δεδομένο όσον αφορά τι Τρίτον, οι προδιαγραφές στην εσωτερική αγορά θα εναρμονίσουν και πρακτικές. όπως το θέμα της ε, οργάνωσης και του εφοδιασμού, τώρα ψηφιοποίηση. Θα είμαι λακωνικός. Θα αναφερθώ σε τρία στοιχεία. Η βιομηχανική ψηφιοποίηση και η σχετική στρατηγική προέρχεται από την έκθεση της ΣΥΤΡΕ που προτείνει στατική συντονισμού της διαδικασίας ψηφιοποίησης και αν είναι πραγματική στρατηγική και υλοποιηθεί θα είναι υποφελής για τις μεταφορές. Εκεί χρειάζεται πράγματι μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ των τομέων και των δύο επιτροπών που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Μετά, επενδύσεις για καινοτομία, για υποδομές, για να γίνει μετάβαση σε ψηφιακές διαδικασίες που απαιτούν επενδύσεις. Αν δούμε το ΕΦΣΙ, που ήδη αναφέρθηκε, σε διαφορετικό πλαίσιο βέβαια, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι σημαντικός φορέας που οδηγεί σε προστιθέμενη αξία. Και αναφέρθηκε και το θέμα του σωστού σχεδιασμού. Αν δούμε σήμερα το πώς τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι θέμα προσωπικό. Μπορεί κάποιοι να είναι ικανοποιημένοι με το ΕΦΣΙ μέχρι τώρα για καινοτόμα προγράμματα. Εγώ είμαι Τσέχος και δεν είμαι ικανοποιημένος. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να βελτιωθούμε και το ΕΦΣΙ μπορεί να παίξει σημαντικότατο, ζωτικό ρόλο στις προσπάθειές μας. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό που λέω. Τα αυτόματα αυτοκίνητα. Ενδιαφέρον Πολύ ενδιαφέρον. Θα μ' άρεσε. Δεν λέω ότι δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για κάτι τέτοιο. Αν δείτε την ανακοίνωση όμως, φαίνεται σαν να είναι ο ακρογωνίος λήθος. Το θέμα. Αυτό που λείπει είναι ότι δεν τονίζεται παρκώς άλλη πτυχή, άλλα έργα, άλλες προπτικές, άλλοι τομείς εκεί που μπορούμε να έχουμε πιο πολύ άμεσα αποτελέσματα, πιο άμεσα αποτελέσματα. Το θέμα ασφαλείας και λοιπά συμφορήσεως στους δρόμους, όταν εξετάζουμε σε σχέση με το όλο περιβάλλον, πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί στην προσέγγιση. Όχι καινοτόμοι τόσο, όσο δημιουργικοί. Μπαίνοντα στι λεπτομέρειε τι βλέπουμε. Ότι κάποιοι από του άλλου τομεί μπορεί να μας οδηγήσουν στα αυτόματα αυτοκίνητα. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Θα ήθελα να εστιαστούμε όχι το κατά πόσο και τι, αλλά το πώς πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να μας βοηθήσουν να κινηθούμε αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τώρα Έχω το λόγο, δίνω το λόγο στον κύριο Καπ και σε στους υπόλοιπους που εκπροσωπούν πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ ε, πραγματικά θερμά τον εισηγητή για όλη τη, δουλειά που έκανε. Δυστυχώς η κυρία Βελκούν δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα. Μου ζήτησε λοιπόν να σας πω ποια είναι τα σχόλιά της εκ μέρους του ΕΛΚ και γενικότερα πρέπει να σας πω πως συμφωνούμε με τα όσα έχει προτείνει και στις διογνωμοδοτήσεις ο συνάδελφος και για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας αλλά και στη γνωμοδότηση για τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να σας πω πώς μπορούμε να συζητήσουμε όλες τις υπέροχες νέες ιδέες που γεννιούνται. Το ζήτημα είναι το πώς θα τις εφαρμόσουμε. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή καταρχήν. Πού βρισκόμαστε σήμερα, έχουμε κάνει μια απογραφή της κατάστασης στην Ευρώπη. Είμαστε ακόμα μπροστά, πώς αντιμετωπίζουμε την Κίνα, την Ινδία, γιατί ξέρετε πως οι δικές τους βιομηχανίες ε, σπέβδουν ταχύτατα ε, προς την ψηφιοποίηση και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που συζήτησε η Ήτρε μήπως θα έπρεπε να μας δώσετε πιο πολλά στοιχεία και όχι απλώς ένα κατάλογο αγαθών προθέσεων. Μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είδαμε τι γίνεται με πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις. Στη ΣΥΠΑ για παράδειγμα και στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις αυτές είναι πραγματικά φρέσκες και ε, καινοτόμες ε, στην ψηφοποι... στο θέμα της ψηφιοποίησης. Άρα λοιπόν η Ήτρε μήπως θα έπρεπε να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές και με ποιο τρόπο. Ο εισηγητής λέει πως έχουμε υποεκτιμήσει τον κλάδο του τουρισμού. Πρέπει να σας πω πως εγώ χρησιμοποιήσει το booking ε, στο Άμστερνταμ και πραγματικά με εντυπωσίασε το πόσο πετυχημένη είναι αυτή η πλατφόρμα. Νομίζω ότι είναι ε, τρομακτικό, είναι τεράστιο, τεράστια βιομηχανία τώρα ο ψηφιακός τουρισμός και νομίζω ότι το δυναμικό εκεί ε, είναι απίστευτο και θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση τώρα για το θέμα των προτύπων και τη δήλωση του Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια της ε, Ολλανδικής Προεδρίας πρέπει να σας πω πως μιλήσαμε για τα αυτόματα αυτοκίνητα, για τα διασυνδεδεμένα, για τα διαλειτουργικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμπεριληφθεί τελικά ε, στην έκθεση και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο αυτή τη δήλωση του Άμστερνταμ. αρμόνιση στην Ευρώπη. Τεράστια επιτυχία. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο μέχρι να επιτευχθεί. Η δική μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξή. Η διαδικασία αυτή είναι θετική. Ποιο έχει καταβάλει το αντίτιμο. Αυτά ήταν λοιπόν τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω στο τραπέζι προ συζήτηση. Merci, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ουζέλη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ταλίτσκα για την γνωμοδότηση που ετοίμασε. Συμφωνώ με τα όσα είπαμε στις βασικές συνομιλίες και εγώ περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει στο μέλλον και για μένα που είμαι Ευρωπαίος πολίτης και για την Ευρώπη. Δεν μιλάω μόνο για την ε, ψηφιοποίηση που αυτή καθεαυτή είναι ένας νέος τομέας που ανοίγεται για τη βιομηχανία αλλά εδώ πρόκειται περί κοινωνιοοικονομικής αλλαγής Πολλοί θα χάσουν τη δουλειά τους και κάποιοι τομείς ε, θα ε, σταματήσουν τις βιομηχανίες. Και έχουμε σαν καθήκον να είμαστε όλοι έτοιμοι σε όλες τις χώρες γι' αυτό και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες διότι θα δούμε αλλαγές μεγάλες τις επόμενες δεκαετίες. Δεν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε με επιτυχία τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή εάν δεν καλύπτεται η διαφορά μεταξύ των πρωτευουσών και της υπαίθρου. Πρέπει να μειωθεί αυτή η διαφορά μεταξύ των διαφόρων περιφερειών για να είμαστε επιτυχείς. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό και για άλλους τομείς όπως είναι αθλητισμός και ο τουρισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις χώρες όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Τι γίνεται όμως με τα μεγάλα δίκτυα που θα ενταχθούν. Η έκθεση αναφέρεται σε αυτά. Όλα τα δίκτυα θα πρέπει να καλύπτονται. Μιλάμε πολύ για το νοδικό τομέα. Αναφερόμαστε στα οχήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους και με τα δίκτυα τα οχήματα που δεν θα χρειάζεται οδηγό. Όμως αυτό θα ισχύσει στο μέλλον, δεν ισχύει σήμερα. Είναι κάτι πολύ απόμακρο σαν προπτική σήμερα. Η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη δεν θα δώσει καρπούς παρά μόνο αν χρησιμοποιήσουμε τις παρούσες τεχνολογίες όπως για την ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και θα πρέπει να πω ότι η ρομποτική είναι ένα θέμα άκρως ενδιαφέρον. Αν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει το ρυθμό, να ανταποκριθεί στο ρυθμό των Αμερικανών και της Κίνας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, να δαπανίσουμε πολύ χρόνο και χρήμα στον τομέα. Όσον αφορά τον τουρισμό, για τον τουρισμό, εκεί όπως είπε ο κ. Βαντεκάμπ στην παρέμβασή του, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο πληροφορικής και σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να αναφερθούμε και στις μεγάλες δημιουργικές βιομηχανίες όπως η εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις έχει μεγάλο μέλλον. Πρέπει να γίνουν τεράστιες ε, επενδύσεις η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν μαζί, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των εργαζομένων και των καταναλωτών. Παραλλήλως, η έκθεση Τελίτσκα ακολουθεί προσέγγιση από πλευρά καταναλωτού. Ίσως θα άξιζε τον κόπο να ακολουθηθεί μια διαφορετική προσέγγιση, μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τους εργαζομένους και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Χρειαζόμαστε σαφείς προδιαγραφές που να μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα σε ένα διεθνές περιβάλλον και που θα επιτρέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ε, διοίκηση την ηλεκτρονική. Χρειάζονται ταχυγράφοι, ταχογράφοι και ηλεκτρονικά διόδια θα έχουμε από πλευρά σοσιαλιστών σχετικές τροπολογίες. Και ευχαριστώ τον κύριο Ταλίτσκα για την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιλόνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Yhtä mieltä äh, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμφωνήσει κανείς με τον εισηγητή του θέματος. Η τυποποίηση και η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε ε, σε αυτή τη φάση. Και θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την τυποποίηση. Αν δούμε λιγάκι την τυποποίηση θα πρέπει να ισχύει για την συγκράτηση και την διάδοση των πληροφοριών και το ρόλο που μπορεί να παίξει η πληροφορία στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Υπάρχουν όλο και περισσότερα apps και εφαρμογές Άρα θα πρέπει να υπάρχει η διαλειτουργικότητα των interface ε, και των ε, τραπεζών δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βελτιώσουμε την υποδομή και να δημιουργήσουμε και κίνητρα για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ποια είναι η άποψή μου για μια έκθεση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά επίκαιρη. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία ε, πραγματικά χωρίς προηγούμενο ψηφιακή επανάσταση και θα πρέπει την ε, ψηφιοποίηση να τη δούμε και ως ευκαιρία αλλά και ως παράγοντα κινδύνου γιατί βεβαίως πάντα τα δύο αυτά συνυπάρχουν και νομίζω πως εσείς κύριε Σιγητά μιλήσατε για τις ευκαιρίες που προσφέρει. Ναι, Σίγουρα τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγού είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αλλά θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το θέμα της επαναβιομηχανοποίησης της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Γιατί βέβαια θα πρέπει εμείς να παρακολουθήσουμε έτσι ώστε να μην έχουμε μια αποβιομηχάνηση βιομηχανοποίηση του κλάδου και να δούμε και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτά τα οχήματα χωρίς οδηγό να είναι απολύτως ασφαλή. Έχουμε εναλλακτικά ε, σχήματα, όπως για παράδειγμα τα ατομικά οχήματα, ε, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά είναι κάτι το εκπληκτικό. Τώρα, με την ψηφιοποίηση έχουμε το θέμα που προκύπτει, που είναι η προστασία των δεδομένων. Δεν είναι αμεληταίο. Και είναι ένα θέμα που γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Δηλαδή, ψηφιοποίηση, ναι, Ωραία, αλλά μπορεί εμείς οι ίδιοι οι νομοθέτες να πρέπει καταρχήν όπως είπε ο κύριος Βάντερ Κάμπ πως θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να εμφανιστούν κάποιοι νέοι δημιουργοί, νέοι εφευρέτες, νέες νεοφυείς επιχειρήσεις και να τους στηρίξουμε και να δούμε παράλληλα πώς μπορούμε να βρούμε τις επενδύσεις οι οποίες θα συνοδεύσουν αυτή τη δημιουργικότητα. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Και επίσης να σας πω πως εδώ μιλάμε για έκθεση πρωτοβουλίας σε κάθε περίπτωση και νομίζω πως για το θέμα αυτό, για τα οχήματα χωρίς οδηγό για παράδειγμα, θα μου πείτε πως δεν κυκλοφορεί ακόμα στους δρόμους, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Προσέξτε, ήδη υπάρχουν γιατί αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Εντάξει, δεν έχουμε έγκριση τύπου ακόμα, δεν έχουμε ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, αλλά υπάρχουν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει και στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι κι αλλιώς. Έχουμε την κυρία Ντιπρέ από την DG Move και από την DG Grow. Έχουμε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Έχετε το λόγο λοιπόν και οι δύο. Ne vous disputez Μην τσακώνεστε. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και οι δύο το λόγο. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Δεν σας είχα δει, με συγχωρείτε. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς. Λοιπόν, εξακολουθώ να θεωρώ ότι είμαι και εγώ ο μέλος αυτής της ομάδας τη Επιτροπή, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να έχω πεταχθεί απ' έξω. Τέλο πάντων, η ψηφιοποίηση, κοιτάξτε του κινδύνου, του βλέπω και εγώ να υπάρχουν. Ε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ε, η ιδέα είναι η εξή. Σαν να έχουμε έναν οδηγό που να οδηγεί ταυτόχρονα τρία φορτηγά. Χρήσιμο αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και ο οδηγός ε, ενός αυτοκινήτου και αυτό μας ε, προκαλεί φόβο. Εγώ είμαι εραστής ε, των ράλι, έχω δύο αυτοκίνητα κούρσας αλλά θέλω να οδηγώ μόνος μου. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Αν και η εξέλιξη είναι προς τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τα αυτόματα αυτοκίνητα, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να ε, διαφυλάσσουμε τα χόμπι μας. Και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ε, ένα σύλλογο των εραστών της Αντίκας, ε, αυτοκινήτων Αντίκας, και για το αυτοκίνητα κούρσα. Στο μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να ασχολούμαστε με το χόμπι μας. Υπάρχουν και θετικά πράγματα βεβαίως και υπάρχουν κίνδυνοι. Εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα διάφορα συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Ελπίζω η Επιτροπή και οι διάφορες διευθύνσει να συμφώνησαν μεταξύ τους, ε, γιατί καταλαβαίνω βέβαια πως χάρη ναυρότητα θέλετε να ξεκινήσει ο άλλο, αλλά πρέπει κάποιος να μιλήσει. Είμαι από την Digiconnect, εγώ. Okay. So, and, and I would just like to... Είμαι από την Digiconnect, Connect εγώ. Και θα ήθελα να μιλήσω για την ψηφιοποίηση της ε, βιομηχανία και σε ευχαριστώ πολύ για τα τόσο πολύτιμα σχόλιά σα, με τα οποία εμείς θα συμφωνήσουμε. Θα ήθελα απλώ να αναφερθώ στο εξή. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του κλάδου των μεταφορών ευρύτερα. Όπω επίση και για το γεγονό ότι αλλάζουν οι κανόνε του παιχνιδιού ε, με την ψηφιοποίηση. Εσεί μιλήσατε για την χρήση δικτύων 5G στην περίπτωση αυτή και υπάρχουν και άλλα εμπόδια στην περίπτωση αυτή τη διασυνδεσιμότητα. Τώρα για τον βιομηχανία επικοινωνία στην Ευρώπη, ξέρετε πω με τον τρόπο αυτό θα συνδεθούν όλοι οι κλάδοι, όλε οι εταιρείε, όλη η βιομηχανία, ανεξάρτητα μεγέθου, ανεξάρτητα τοποθεσία, θα έχουν την πρόσβαση αυτή στην ψηφιακή τεχνολογία και στι ε, δεξιότητε έτσι ώστε να περάσουν σε αυτή τη μεταψηφιακή εποχή. Και δώσαμε συγκεκριμένα προβλήματα όπου οικοδομώντας αυτές τις ψηφιακές βιομηχανικές πλατφόρμες θα προωθήσουμε με πολύ καλό τρόπο την αντιγυνιστικότητα της Ευρώπης. Και έτσι δεν θα έχουμε μόνο ε, το θέμα των οχημάτων χωρίς οδικό, ε, οδηγό ή ε, των διασυνδεδεμένων οχημάτων. Όχι, θα είναι πολλά ακόμα. Τώρα, εδώ, σε αυτά τα παραδείγματα, ναι, όντως, για μεγάλα πειραματικά έργα έχουν διαθέσει πάρα πολλά κονδύλια σε όλη την Ευρώπη, αλλά εκτός από το θέμα αυτό, έχουμε την διαχείριση κυκλοφορίας πληροφορίας ε, την συγκοινωνία και τις πληροφορίες ε, για τα μέσα μαζικών συγκοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και άλλα πολλά ακόμα. Και ξέρω πως ο συνάδελφος, για παράδειγμα, από την DG Move μπορεί να σας πει παραπάνω. Εγώ θα ήθελα μόνο να ρωτήσω το εξής. Το ΕΛΚ λέει πως η διαδικασία ψηφιοποίησης δεν ήταν σε όλο, για τον όλο τον κλάδο των μεταφορών εξίσου ευνοϊκή. Θα ήθελα εδώ να μου πείτε κάτι παραπάνω. Τι ακριβώς έχετε κατά νου. Δίνω το λόγο τώρα στους συναδέλφους. Δεν είναι η κυρία Ντεπρέ, έκανα λάθος. Η κυρία Βαντόμ, ε? Από την Τζιμού, βορίστε, έχετε το λόγο. Μιλήστε. Ευχαριστώ πολύ, Ισαμπέλ Βαντεμπορν. Είμαι ένα βοηθός της κυρίας Ντεπρέ. Στην στη DigiMove ε, με τα χαράς ε, είδαμε το σχέδιο γνωμοδότησης διότι πάντα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας ο μεταφορικός και στο εγγύς και στο μακρινό μέλλον. Για το εγγύς ή το απόμακρο μέλλον δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση υπάρχει, είναι εδώ και πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οπότε συμφωνούμε με αυτά που είπε ο συνάδελφο τη DG Connect σχετικά με την ψηφιοποίηση. Και επεξεργαζόμεθα τα διάφορα θυγέντα ζητήματα. Τώρα, αν θέλετε να μπούμε σε λεπτομέρειε, υπάρχει οριζόντια προσέγγιση, όπως αυτή που ακολουθείτε με την ανακοίνωση για την οικονομία των δεδομένων. Υπάρχει και άλλη οδηγία, η οδηγία PSI Directive. Επίσης έχουμε και τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Όλες αυτές οι οριζόντιες εργασίες ισχύουν και για τις μεταφορές. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ακόμα σημεία προσκάλυψη για τις μεταφορές να επανεξεργαστούμε οριζοντίως το θέμα και μετά να απαιτείται βλέπουμε αν υπάρχουν ειδικά σημεία που αφορούν τις μεταφορές, σε πάση περιπτώσει. Το σχέδιο γνωμοδότησης το στηρίζουμε. Είναι πολύ καλό κατά την απόψή μας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξανά το λόγο τον έχει ο εισηγητής. Για να ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι γρήγορος. Ε, θα αναφερθώ στα σχόλια των συναδέλφων και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Βαντεκάμπ, που βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Υποκειμενικό ερώτημα, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Αν κρίνω βάσει δικών μου κριτηρίων, θα έλεγα ότι δεν είμαστε τόσο μπροστά όσο θα μπορούσαμε. Αναφέρθηκε στη συζήτηση άλλωστε από κάποιες πτυχές, κάποιες χώρες, είτε είναι η Κίνα, σε άλλα στοιχεία, άλλες χώρες είναι πιο μπροστά. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχουμε μία λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Είναι η αγορά. Σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε. Αν εξαρτάται αυτό από τους ε, κανόνες, το ρυθμιστικό περιβάλλον και την εποπτεία, είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Κίνα. Χρειάζεται ένας ρυθμιστικός φορέας. Και όχι στην Ευρώπη είναι διαφορετικό. Έχουμε 28 συν 1. Δεν είναι κακά τα πράγματα, δεν είναι δραματικά αλλά βλέπουμε ότι και με τις επενδύσεις που γίνονται σε άλλα σημεία του πλανήτη γίνονται τεράστιες επενδύσεις. Πολλοί δικοί μας που είναι έξοχοι όσον αφορά την καινοτομία στο ψηφιακό τομέα και στις μεταφορές τους βλέπουμε στη Silicon Valley. Γιατί? Διότι υπάρχει κεφάλαιο εκεί και δεν ε, έχουμε στην Ευρώπη. Ε, όχι, καθόμαστε το κεφάλαιο, έχουμε πολύ. Αλλά θεωρούν ότι είναι πιο ελκυστικό να πάνε στις Ηνωμένες όχι σε κάθε τομέα, υποτομέα, αλλά αποτελεί πρόβλημα αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματική ενιαία αγορά και κάποιος αναφέρθηκε και στα κίνητρα. Τώρα όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις, συμφωνώ. Μπορούμε να το εξετάσουμε, να δούμε αν μπορούμε να το τονίσουμε περαιτέρω. Εγώ υποστηρίζω ένθερμα τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι, την ψηφιακή εποχή, σε αυτό το τομέα οι νεοφυείς επιχειρήσεις κυρίως είναι η κινητήρια δύναμη. Και να δούμε τι κίνητρα μπορούμε να τους δώσουμε στο μέλλον. Τυποποίηση, εναρμόνιση, αν είναι θετικό αυτό, εν γέννη είναι θετικό. Εξαρτάται πώς γίνεται η τυποποίηση. Μπορεί να κάνει κανείς και λάθη, αλλά εν είναι. Ο κύριος Γιέλη για τους σοσιαλιστές ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στους κινδύνους Αναφέρθηκε και στους εργαζομένους. Είπατε υποβάλλετε σχετική τροπολογία. Εγώ είμαι υπέρ. Αλλά θα ήθελα να αποφύγουμε την εξή περίπτωση. Σαν Επιτροπή Μεταφορών, αμέσως γνωμοδοτήσεως ή εκθέσεως, ετοιμάζουμε έκθεση που αφορά μία πλευρά της εργοδοσίας. Εγώ είχα την εμπειρία από τις αερομεταφορές. Ήταν ένας εφιάλτης η κατάσταση βάσει όσων είπατε δεν έχω πρόβλημα με τα χαράς να δω την τροπολογία σας. Και μπορούμε να βρούμε διέξοδο. Έγινε λόγος ε, για τον τουρισμό. Το ανέφερε και ο κ. Κάμπ. Και εδώ καλά τα πάμε. Αρκετά καλά. Αναφερθήκατε στην Booking.com θα ήθελα εδώ τη μέρα όμως που μπορώ να καθίσω στον υπολογιστή μου και μέσω της Booking.com να μην κλείσω μόνο ξενοδοχείο, αλλά να βγάλω και εισιτήρια μέσω διαφόρων μέσων να φτάσω στο ξενοδοχείο που θα μείνω. Όλοι ξέρουμε ποια είναι τα εμπόδια. Και ρητορικό είναι το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά τα προβλήματα και τις συμφορήσεις. Τώρα, ποιε είναι οι συνέπειε για του εργαζομένου από τη ρομποτοποίηση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πήγαμε στη Χιλή Δημοκρατία σαν Επιτροπή Μεταφορών και πήγαμε σε μια εγκατάσταση με οδηγό που χρησιμοποιούσε όχημα που ήταν ημιαυτόματο, παρόλα αυτά ήταν παρόν ο οδηγό, Κάθε βιομηχανική επανάσταση έχει αντίκτυπο. Όχι μόνο για την εργοδοσία και την απασχόληση, αλλά για τη φύση της εργασίας επίσης, την ποιότητα της εργασίας. Και είναι μια διαδικασία η οποία θα κάνει τι προσαρμογέ τη. Όσον αφορά την κοινή χρήση υποδομών και κίνητρα. Α, έφυγε ο συνάδελφος που έθεσε το θέμα. Καλό αυτό όμως. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι αμέλησα το ότι έρχεται ο αυτοματισμός. Όχι, όχι, όχι, παρεξήγηση είναι. Είπα κάτι διαφορετικό. Κάτι στο οποίο απάντησε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ότι εστεζόμεθα σε κάτι πολύ ελκυστικό, στα αυτόματα αυτοκίνητα σήμερα. Αλλά έχουμε πολλού άλλου τομεί και προπτικέ που έχουν δρομολογηθεί. Μπορούμε να συζητούμε εκεί. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα, είναι πιο άμεσα τα αποτελέσματα αναμενόμενα. Αλλά εγώ είμαι ο τελευταίο που θα έλεγα ας περιμένουμε, διότι δεν είναι πραγματικότητα αυτόματα αυτοκίνητα, ας περιμένουμε τον κανονισμό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την ημέρα που από τη στιγμή το αυτοκίνητο παρκάρει μόνο του τώρα στο μέλλον που θα έχουμε πλήρω αυτοκίνητο που θα είναι πλήρω αυτόματο και θα σε πηγαίνει στον προορισμό σου. Η προστασία των δεδομένων εξυπακούεται. στον ψηφιακό τομέα, είτε στις μεταφορές, είτε και σε άλλους τομείς. Ο κύριος Λούγκρεντ. Σας κατανοώ. Σας καταλαβαίνω. Και, εγώ, και εμένα μου αρέσει η οδήγηση. Όπως σας είπα, δεν θα έρθει και τόσο γρήγορα αυτό. Θα πρέπει όμως να αλλάξουμε και εμείς σχολείες και χόμπι. Αλλάζει ο κόσμος. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελικά σχόλια. Είπατε ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι εποφελής για κάθε τρόπο μεταφορών. Όχι. Στους σιδηροδρόμους έχει το ERTMS ενώ αν θέλω να κινηθώ διασυνοριακά αν διαστήσεις τέσσερις χώρες πρέπει να αγοράσεις αυτοκόλλητο μια βινιέτα σε κάθε σύνορο και να το κολλάς για να προχωρήσει. Αυτό είναι ένα παράλογο παράδειγμα. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα διαφορετική κατάσταση στις αερομεταφορές από τις οδικές. Έχουμε μείνει πολύ πίσω στις οδικές. Αν δείτε στο μεταφορά φορτίων, εκεί υπάρχει βελτιστοποίηση όσον αφορά τη χρήση των οχημάτων, υπάρχει λογισμικό, ψηφιοποίηση κλπ. Όσον αφορά μεταφορά επιβατών, ναι, έχω ψηφιακό πίνακα που μου λένε ότι κάπου συνέβη ένα τύχημα στα 3 χιλιόμετρα από εδώ. Υπάρχει τεράστια διαφορά όμως, ε. Ε, σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο ετοιμάζουμε το ρυθμιστικό περιβάλλον. Κυρία Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαντεκάμπ, θέλετε να χειροκροτήσετε. Εκτός μικροφώνου απάντηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλη σας τη δουλειά κύριε Σίγητα. Νομίζω ότι τελειώσαμε ε, για σήμερα. Αύριο το πρωί θα τα πούμε πολύ νωρίς και θα μείνω εδώ μόνο με τους εισηγητές, μια και θα είμαστε ε, και κλεισμένων των θυρών. Οι συντονιστές μόνον και σας υπενθυμίζω πως οι τροπολογίες για την έκθεση Τελίτσκα και για τα δύο θέματα είναι η 6η Μαρτίου του μεσημέρι. Κάνουμε λοιπόν πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές μόνον. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, πρωί-πρωί στις 9.